Dear colleagues, good afternoon. We can continue our program by point number 25. Καλησπέρα, μπορούμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το σημείο 25, ανταλλαγή απόψεων για με την κυρία Λουτσία Ζήτνιανσκα, αντιπρόεδρος και υπουργός ε, ε, Δικαιοσύνης της Σλοβακίας και ο κύριος Ιβάν Τσέντσης, ε, Υπουργός ε, Πολιτισμού και θα μας κάνει μια ενημέρωση για τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας. Έχουμε οργανώσει το σημείο αυτό έτσι ώστε να κάνουμε μια εισαγωγική παρουσίαση ο καθένας από τους προσκεκλημένους του μας και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τους υποβάλουμε ερωτήσεις και στους δύο ταυτόχρονα. Ξεκινάω λοιπόν δίνοντας ε, το λόγο στην ε, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης, κυρία Ζητνιάνσκα. E, Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, Πριν από λίγες μέρες ε, η Σλοβακία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου δίνεται να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Για ε, αυτές που αφορούν ε, τι αρμοδιότητε αυτής εδώ της Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει πολλέ προκλήσει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Στο πλαίσιο αυτό ο τομέας του αστικού δικαίου, της δικαστικής συνεργασίας και του εμπορικού δικαίου ίσως να μην είναι και τα θέματα με την υψηλότερη προτεραιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο άλλα θέματα που συζητώνται εκτενώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι τομείς αυτοί είναι εξίσου σημαντικοί, διότι πολύ συχνά επηρεάζουν άμεσα πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο πολιτών όσο και επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα όσον αφορά τη διασυνοριακή εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Στον τομέα αυτών ε, η Σλοβακική Προεδρία θα ήθελε να προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες τις οποίες μπορούμε να ομοδοποιήσουμε υπό τον τίτλο e-justice, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ε, ειδικότερα ηλεκτρονική επικοινωνία στον τομέα της δικαιοσύνης, που θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου τόσο για αστικές όσο και για εμπορικές υποθέσεις. Ο τομέας αυτός αφορά επίσης και την επίδοση των δικαστικών εγγράφων, την ε, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και επ' αυτού θα διοργανώσει η Σλοβακή Προεδρία μια διάσκεψη στην Πρατισλάβα, στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, ε, τον Οκτώβριο. Η διασκέψη αυτή θα εστιαστεί στην επίδοση δικαστικών εγγράφων και παράλληλα με αυτήν ε, το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστικό Δίκτυο για Εμπορικά και Αστικά ε, θέματα θα λάβει επίσης χώρα. Ελπίζουμε έτσι λοιπόν να προχωρήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν που προβλέπει να αναθεωρήσει τον κανονισμό για την επίδοση των δικαστικών εγγράφων και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Με τι ε, προκλήσει που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δημιουργία μια ενιαίας ψηφιακή αγορά. Στον τομέα αυτόν έχει να σημαντικό ρόλο, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι οδηγίε ή η οδηγία για το δίκαιο των συμβάσεων που ρυθμίζει τις πωλήσει υπηρεσιών και αγαθών. Η Σλοβακική Προεδρία θα συνεχίσει τη συζήτηση η οποία ξεκίνησε με εντατικού ρυθμού κατά τη διάρκεια τη Ολλανδική Προεδρία. Η Ολλανδική Προεδρία επικεντρώθηκε κυρίω στην πρόταση που αφορά το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό περιεχόμενο. Εμείς ε, προβλέπουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, στον τομέα αυτόν. Ε, ελπίζουμε σε μεγάλο βαθμό αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτέ οι δύο προτάσεις ε, σχετίζονται στενά μεταξύ του. και είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε κάποιο συντονισμό, κάποια αρμονία μεταξύ του Γι' αυτό τον λόγο η Σλοβακική Προεδρία προβλέπει να ξεκινήσει μια σημαντική, μια ουσιώδη συζήτηση επί της πρότασης ε, περί επιγραμμικών πωλήσεων μόλις ε, τα πρώτα αποτελέσματα ε, του refit του κεκτημένου για τους καταναλωτές ε, έχουν βρεθούν στα χέρια μας. Εμείς αναμένουμε αυτά τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα το Σεπτέμβριο φέτος. Άλλο ένα θέμα σημαντικό για τη Σλοβακή Προεδρία τουλάχιστον είναι η εκκίνηση των τεχνικών συζητήσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 σημαντικός κανονισμός για το οικογενειακό δίκαιο, για το διεθνές οικογενειακό δίκαιο. Βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και πάνω από 10 χρόνια και η αναθεωρησή του μας δίνει την ευκαιρία να ε, αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Και να εξετάσουμε τα ζητήματα που επισημανθήκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά του έγγραφα. Θέλουμε να εντείνουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να τη βελτιώσουμε. Φυσικά δεν αναμένουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό με το τέλος της Προεδρίας μας, ωστόσο η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλό ανοιχτό περιβάλλον που να λειτουργεί σωστά όπου υψηλού επίπεδου συζητήσει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα είναι δυνατόν να λαβούν χώρα. Κατά τη Σλοβακική Προεδρία το Συμβούλιο θα συνεχίσει την πολιτική του στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες ε, δύναμη της διάσκεψης της ε, Χάγης για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο Όσον αφορά για το δίκαιο εμπορικών εταιριών, η Σλοβακία θα συνεχίσει τις ε, συζητήσεις ε, σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων και συμμεριζόμαστε τους φόβους που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων κατά χώρα. Μετά από ανάλυση και εκτίμηση αντικτύπου, η Κομισιόν υπέβαλε μια νέα πρόταση όπου το country by country reporting, η υποβολή εκθέσεων κατά χώρα, έχει ε, ενσωματωθεί με την ε, οδηγία περιλογιστικής. Φαίνεται να είναι η λύση που αρμόζει για την κατάσταση όπως έχει. Όπως λοιπόν και η προηγούμενη Προεδρία, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε και έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα υπόλοιπα κομμάτια της πρότασης μέχρι ότου το ζήτημα της ε, υποβολής εκθέσεων κατά χώρα επιληθεί ώστε ουσιαστικά όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι έως ότου μείνει ικανοποιημένο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δηλαδή το συγκεκριμένο αυτό ε, στοιχείο δεν εξετάζεται στην οδηγία περί δικαιωμάτων των ε, μετόχων για τη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένη ευθύνη, η Σλοβακή Προεδρία θέλει να επιτύχει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον για το ζήτημα αντιμετώπιση αυτού τη πολύ ευαίσθητη πρόταση στο μέλλον. Επειδή υπάρχει μια τάση απλούστευση τη πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, το Συμβούλιο εμένει ε, ότι η πρόταση αυτή θα ωφελήσει ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο φυσικά είναι έτοιμο να καθησυχάσει οποιασδήποτε ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να λάβει τα σχετικά μέτρα ε, σε σχέση με πιθανή κατάχρηση αυτής της νομικής πράξης ε, για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος ε, και της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στα πλαίσια φυσικά της εργατικής νομοθεσίας. Ξέρω ότι η παρούσα Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης για τα θέματα copyright και τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά δεν εντάσσονται στη δικό μου στη Σλοβακική Δημοκρατία, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υφυπουργό Πολιτισμού για να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά θέλω να σα εκφράσω την πεποίθησή μου ότι κατά τη Σλοβακική Προεδρία η καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου θα φέρει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, στην εισαγωγή μου ξέχασα να τονίσω ότι η κυρία Ζητνιάνσκα βρίσκεται πολύ κοντά στην Επιτροπή μας επειδή είναι καθηγήτρια εταιρικού δικαίου. Οπότε κάνετε τις δύσκολες ερωτήσεις. Γι' αυτό το λόγο. Προτείνω τώρα να ακούσουμε, να μάλλον ερωτήσεις και απαντήσεις ε, μετά από την παρουσίαση του κύριου Ιβάν Σέτσεκ. Αναπληρωτής ε, Υπουργός Πολιτισμού, στον οποίο δίνω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που καλούμε να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη εκ μέρους της Σλοβακικής Προεδρίας και της ε, και του Συμβουλίου. Μια από τι προτεραιότητε τη Προεδρία μα στο Συμβούλιο είναι η υλοποίηση τη στρατηγική για την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά και ο εξυγχρονισμό φυσικά του πλαισίου copyright για τα πνευματικά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη πρωτοβουλία τη Κομισιόν σε αυτό το τομέα ήταν η πρόταση για του κανονισμού για τη φορητότητα των ε, ψηφιακών υπηρεσιών αυτό που ουσιαστικά ονομάζουμε εν συντομία πρόταση για τη φορητότητα. Εδώ καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ολλανδική Προεδρία κατάφερε μέσω τη επικοδομητική προσέγγιση μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, κατάφερε να επιτύχει κάποια αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι μετά από πολύ εντατικέ ε, συζητήσει, κατάφερε το Συμβουλίο να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ε, διασφάλισης της φορητότητας των πόρων μεταξύ χωρών και της ανάγκης ε, ε, να διασφαλιστεί ε, σωστή αμοιβή των δικαιούχων αυτών των δικαιωμάτων. Εμεί θέλουμε να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση, το συντομότερο δυνατόν, διότι πιστεύω θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στου πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, παρότι οι νομοθετικές προτάσεις του δευτέρου πακέτου για το copyright, που δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, η Κομισιόν έχει δημοσίευσει, της, έχει κοινοποίησει στην ανακοίνωσή της ε, προς ένα σύγχρονο πλαίσιο για το κοπηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις προθέσεις της. Και στόχος της Σλοβακικής Προεδρίας είναι να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο στη συζήτηση στο Συμβούλιο, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή οι συζητήσεις αυτές και η όλη μεταρρύθμιση είναι ιδιαίτερα τεχνικές, ε, ε, δεν θα είναι κάτι εύκολο τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright, ε, παίζει σημαντικό ρόλο. Πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδης ε, λήθος, ε, ακρογωνιές λήθος της οικονομίας γνώσης, διότι η γνώση και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι σημαντική για την οικονομία που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό τα πνευματικά δικαιώματα να μην αποτελούν πρόσκομα στην ανάπτυξη αυτών των στοιχείων της γνώσης και της πρόσβασης της πληροφορίας. θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές ε, στο νομοθεσία του copyright. Διότι πιστεύουμε ότι αυτή η νομοθεσία για τα πραγματικά δικαιώματα θα είναι κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη των επωνομαζόμενων βάσεων δεδομένων μνήμης που συνοψίζουν ουσιαστικά τις γνώσεις μας. Τώρα, η έλευση των νέων ε, ψηφιακών τεχνολογιών, αυτό είναι ένας άλλος τομέας. Ε, θα μας επιτρέψουν αυτές οι νέε τεχνολογίε να αξιοποιήσουμε τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και το ψηφιακό περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να άρουμε οποιαδήποτε εμπόδια μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού κόσμου και να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχή των νέων ψηφιακών υπηρεσιών, του νέου περιεχομένου. Σήμερα, στο ψηφιακό περιβάλλον, οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας άλλων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ανταμείβονται με διαφανή και δίκαιο τρόπο και η όχι των δικαιωμάτων αυτών. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των δικαιούχων ε, ε, των δικαιωμάτων αυτών. Η Σλοβακική Προεδρία πιστεύει επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να εστιαστούμε στη διαδικασία της επικύρωσης της ε, Συμφωνίας του Μαρακές που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε περιεχόμενο για ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης. Πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να διασφαλίζονται μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στα διάφορα έργα και στα αντίτυπά τους ε, με προσπελάσιμες ε, μορφές ε, με δυνατότητα πρόσβασης από οποιουσδήποτε συμβαλόμενος και νομικά πρόσωπα. Και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν ακόμα όσον αφορά την εντολή για την επικύρωση και όσον αφορά και την νομική βάση. Εμείς πιστεύουμε ότι μετά από την γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί μια λύση. Έτσι ελπίζουμε. Γι' αυτό το λόγο η Σλοβακική Προεδρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μόλις το, η γνωμοδότηση του δικαστηρίου δημοσιευτεί. Εκεί θα συζητήσουμε με την Κομισιόν και θα προχωρήσουμε το θέμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ωραία, αγαπητοί συναδέλφοι. Μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Ε, έχω μία πολύ σύντομη ερώτηση να σας υποβάλω ε, προς εσάς, κυρία Σινιάτσκα. Συγκεκριμένα πρόκειται για το εξή. Βεβαίω μας καθησυχάζει πάρα πολύ το ότι μια καθηγήτρια για το εταιρικό δίκαιο, δηλαδή για θέματα που είναι σημαντικά, όπω οι εκτέσει αναχώρα, ότι για το θέμα αυτό ε, ασχολείται μία κατηγήτρια. Και επίση είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι η Σλοβακική Προεδρία θα προσπαθήσει να προωθήσει το θέμα αυτό. Αλλά η ερώτησή μου αφορά ένα άλλο θέμα, ένα θέμα για το οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πρόκειται για τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers όπως λέγονται. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και έχει άμεση σχέση με το εταιρικό δίκαιο, δηλαδή ε, όλα αυτά που διαρρέουν ε, διάφορες περιπτώσεις, τελευταία τα Panama Papers, είναι θέματα που απασχολούν την δική μας την Επιτροπή, την Νομική Επιτροπή. Σας ερωτώ λοιπόν, το θέμα των καταγγελόντων, των whistleblowers, θα το εξετάσετε κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας ή όχι. Η Κομισιόν δεν έχει υποβάλει ακόμα συγκεκριμένη πρόταση, αλλά ο συνάδελφός σας, ε, ο Σλοβάκος ε, στην Ολομέλεια, είπε ότι προτίθεται να ακολουθήσει έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τη Σλοβακική Προεδρία στην Επιτροπή μας και προσβλέπω στην αγαστή συνεργασία. Εγώ είμαι η συγγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, για την επιγραμμική πώληση των ε, ενσώματων αγατών. Νομίζω ότι είπατε κι εσείς ότι προτιμάτε να περιμένετε μέχρι να προκύψουν το Σεπτέμβρη τα αποτελέσματα του REFIT για να τοποθετηθείτε επί της πρότασης της Επιτροπής. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, διότι στο Κοινοβούλιο σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες θα επιθυμούσαν διακαώς αυτή τη δουλειά ε, για τα ενσώματα αγατά να ευθυγραμμίζεται η δουλειά με την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά θέματα ε, τα οποία πρέπει κανείς να εξετάσει, ενδεχομένως το θέμα της ευθυγράμμισης. δεν ξέρω, το Συμβούλιο θα περιμένει μέχρι το Σεπτέμβρη για τα ενσώματα αγατά. Αν είναι έτσι, τότε το πρόγραμμά μας που λέει να δουλέψουμε γρήγορα, μάλλον δεν βγαίνει. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, τι προτίθεστε να κάνετε για να προχωρήσετε και πιο γρήγορα όλη αυτή η δουλειά που γίνεται για τα ενσώματα αγαθά. Ε, ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στη Σλοβακική Προεδρία γιατί ξέρετε τα έχετε αντιμετωπίσετε δύσκολα θέματα. Επειδή έρχομαι από τη Ρουμανία Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον προτίθεστε να συζητήσετε για τη διεύρυνση του Σανκέν με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Εγώ μιλάω πρώτα για τη Ρουμανία, γιατί ξέρετε καθαρά τεχνικά η Ρουμανία καλύπτει όλα τα τεχνικά προαπαιτούμενα για να ενταχθεί στο Σανκέν. Επιπλέον η Ρουμανία προσφέρει ε, σταθερότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και δεν καταλαβαίνουμε. Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί η αρμόδια αρμόδιοι αρνούνται να δεχτούν τη Ρουμανία στο Σέγγεν. Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή είσαστε επαΐουσα στο εταιρικό δίκαιο, αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει εισάγει τον κατώτατο μισθό για τους οδηγούς φορτηγών. Ακόμα και για αυτούς ε, που προέρχονται, ε, που διασχίζουν τη χώρα ε, με τη μορφή τράνζιτ. Το ίδιο σκοπεύει να κάνει και η Γαλλία. Εσείς τι πιστεύετε για το θέμα αυτό. Και η τελευταία μου ερώτηση σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων. Τι έχετε να προτείνετε μετά από τις 16 ώρες πρέπει να υπάρχει κάποια πάψη. Τι ε, ε, σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα των εργαζομένων, γιατί έχει ήδη προταθεί το θέμα της κίτρινης κάρτας. Πρόεδρος, ε, πρέπει να σας πω όμως ότι η κυρία Ζουσάτκα δεν είναι υπουργό εσωτερικών, άρα δηλαδή αυτό που ρωτήσατε για το Σέγκεν ε, δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές της. Ο κύριος Κοφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θέλω λιγάκι να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο παρουσιάσατε σε σχέση με τις συστάσεις, τις εκθέσεις μάλλον, εκθέσεις αναχώρα. Ισχύει το εξής. Εμείς ε, αυτό το συζητήσαμε και στην Ολομέλεια. Πρόκειται για την οδηγία περί των δικαιωμάτων των μετόχων. Εμείς ε, συζητήσαμε για αυτή την οδηγία, διεξοδικά μάλιστα, ε, κατά διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Σημειώθηκε αρκετή πρόοδος και θέλουμε κάπως με τη δική σας τη βοήθεια να κλείσει το θέμα. Και θα με ενδιαφέρει λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσον και εσείς ενδιαφέρεστε για το ίδιο πράγμα. Και θέλω να προσθέσω ότι αν τελικά μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα θέμα που να είναι λίγο πολύ, πολύ κοντά στο τέλος της οδηγίας, να τελειώνει δηλαδή αυτή η οδηγία για τους ε, μετόχους, αυτό θα βοηθούσε στο να ολοκληρωθεί και η οδηγία των εκθέσεων αναχώρα. Άρα δηλαδή νομίζω, κατά δική μου άποψη, είναι πολύ σημαντικό το τι στάση θα κρατήσετε εσείς σε αυτή την οδηγία για τους ε, μετόχους και επίσης ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κατά πόσον θα επιταχύνεται ε, όλη αυτή την υπόθεση των ε, εκθέσεων αναχώρων γιατί και τα δύο πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Αλλά όσο πιο γρήγορα προχωρήσετε για το ένα θέμα, τόσο πολύ πιο εύκολα θα είναι να λυθεί και το άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Σβεύκα. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα... Ε, να ρωτήσω, ε, να απευθυνθώ στον κύριο Ναπληρωτή Υπουργό. Ε, χαιρόμαστε που ήρθατε και ε, χαιρόμαστε που ακούσαμε το τι προτίθεστε να κάνετε τους επόμενους έξι μήνες. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μισό χρόνο. Για μας βέβαια τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα γιατί από τους έξι μήνες θα χαθούν οι δύο. Πάει ο Ιούλιος, πάει και ο Αύγουστος. φτάσαμε στο Σεπτέμβριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, θα είσαστε η προεδρεύουσα χώρα και χαίρομαι που θέλετε να προχωρήσετε τα θέματα και δεν λέτε ότι αυτό το θέμα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει υπό την Προεδρία μας. Γιατί αυτό το κάνουν ε, συχνά πολλές Προεδρίες και ξέρετε τι γίνεται. Τελικά αυτά που έχουν ανακοινωθεί δεν ολοκληρώνονται. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο στόχος σας ε, που είναι να είσαστε πιο επικοινωνιακοί, να λειτουργούν καλύτερα τα θέματα. Αυτό είναι καλύτερο και είναι πολύ πιο σημαντικό το ότι δεν μπαίνετε τόσο στα νομοθετική φύσεως θέματα. Εγώ λοιπόν είμαι εισηγητή που αφορά στην επεξεργασία του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Χθε είχαμε ανταλλαγή απόψεων, πολύ ενδιαφέρουσα, με εκπροσώπους της Επιτροπής και εκεί κατέστη σαφές το θέμα αυτής της αναδιάταξης και εμείς το συνδέουμε αυτό με τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ε, σε διασυνοριακές αποφάσεις, σε πολλές ε, νομοθετικής φύσεως εξελίξεις. Άρα δηλαδή η αναδιάταξη ε, βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε από αυτού και γι' αυτό σας ερωτώ. Και κατά τα άλλα θέλω να ε, ρωτήσω αυτό πρώτα και ο κύριος Κοφεράτη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί ο διάλογος για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των ε, μετόχων και θα ήθελα να πω για τις εκθέσεις αναχώρα το εξής. Στην τελευταία συνεδρίαση υπό την Ολλανδική Προεδρία διαπιστώσαμε το εξής. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό λοιπόν ε, ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική και ταχεία πρόοδος, να κλείσει σύντομα το θέμα, διότι οι εκπρόσωποι της ε, Σλοβακικής ε, Προεδρίας έχουν συμμετάσχει ενεργά στις ε, τριμερείς συζητήσεις και νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να προχωρήσουμε. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την κυρία Υπουργό και τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό για όλα αυτά που μας είπαν. Τρία θέματα που θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, το επόμενο εξάμεινο ε, υπάρχει η εμπορική συμφωνία ΣΕΤΑ που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Επ' αυτής υπάρχουν πολλές ε, και διαφορετικές νομικές απόψεις για το κατά πόσον θα είναι ένα αμυγός, μια αμυγός ευρωπαϊκή συμφωνία ή θα είναι ε, μια μεικτή συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι νομικά ε, είναι ευρωπαϊκή η συμφωνία, αλλά για καθαρά πολιτικούς λόγους ε, θα πρέπει να συνενέσουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Εσείς τι πιστεύετε από αυτού και πέρα από αυτό έχω και ένα άλλο ερώτημα. Κατά την άποψή σας ε, το διαιτητικό δικαστήριο το οποίο προβλέπεται στη ΣΕΤΑ είναι συμβατό με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν θα έπρεπε καταρχήν να ακούσουμε την άποψη του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν ως Κοινοβούλιο καταλήξουμε σε λάθος άποψη. Καλό που θα προχωρήσουμε στη φορητότητα. Το αναφέρατε το θέμα αυτό και ελπίζω γρήγορα να ε, επιτευχθούν ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Τρίτο θέμα είναι το θέμα δικαιώματα δημιουργού. Και εδώ με ενδιαφέρει το εξής. Ε, στην ψηφιακή ε, βιομηχανία δημιουργών ελοχεύει ο κίνδυνος πλέον οι καλλιτέχνες να μην αμείβονται ικανοποιητικά. Έχετε κάποια ιδέα τι είδους ε, εργαλεία νομικοπολιτικά μπορούμε να εισάγουμε συζήτηση για να διασφαλίσουμε αυτή την ικανοποιητική αποζημίωση των δημιουργών, των καλλιτεχνών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Προφανώς, και το παραλαμβάνω, δεν είμαστε στην Επιτροπή Ιντα, αλλά στην Επιτροπή Γιούρη. Για να είναι σαφές αυτό. Αν όμως ε, θα ήθελε αντιπρόεδρος κυβέρνησης να αναφέρει κάτι σχετικά, ε, μπορεί. Παρακαλώ κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αλλά πρέπει και εγώ να επιβάλλω στον εαυτό μου πειθαρχία για να μην ε, υπερβώ ε, το πεδίο αρμοδιοτήτων και να μιλήσω μόνο για το δικό μου πρωτοφυλάκιο. Καταλαβαίνω την ερώτηση της κυρίας Ρέγνερ. Το θέμα των καταγγελόντων και της προστασίας τους, όπως προείπατε, δεν έχει ακόμη υποβάλει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, θεωρώ ότι το ζήτημα αφορά περισσότερο τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τα εσωτερικά ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, μεν, αλλά σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, εμείς μπορούμε να επεξεργαστούμε μια πρόταση μόνο αφού τη λάβουμε. Επομένω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη πρόταση από πλευρά Κομισιόν, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Και νιώθω και εγώ ότι έχω έναν περιορισμό, ε, λέω υπό κάποιο περιορισμό ως προς αυτό το θέμα. Ε, το δεύτερο ε, που θέλω να πω αφορά ένα ερώτημα του κύριου Ντούντα. Μπούντα. Μιλήσατε για την απόσπαση εργαζομένων, κατώτατο μισθό. Αυτά τα ζητήματα δεν εμπίπτουν ε, στο δικό μου πεδίο αρμοδιοτήτων. Το ερώτημα θα έπρεπε να απευθυνθεί ε, στους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ίδιο ισχύει, το είπε άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κ. Φόποντα, το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τη διεύρυνση του Σέγγεν. Βέβαια εδώ ίσως θα μπορούσα να υπερβώ λίγο το πεδίο αρμοδιοτήτων και να σας διαβιβάσω τις σχετικές πληροφορίες. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ η Σλοβακική Προεδρία ανέφερε ότι θα δρομολογήσει ε, μια συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών για την συμπερίληψη Βουλγαρίας και Ρουμανίας, την ένταξή τους στο χώρο Σέγγεν. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα ερωτήματα που ήταν εκτός δικής μου αρμοδιότητας και τώρα θα περάσω ή μάλλον όχι ακόμη, θα περάσω αργότερα στα δικαιώματα των μετόχων, ε, λίγο πιο διεξοδικά. Πρώτα, μάλλον όχι. Κατευθείαν θα μιλήσω για την οδηγία αυτή. Ε, ε, ε, Πιστεύω ότι αυτή είναι και η άποψη του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά ε, τις εκθέσεις αναχώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό έγγραφο, ένα λογιστικό έγγραφο, ίσως έτσι θα μπορούσε να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Στόχος είναι βέβαια να επιτευχθεί μια, ε, ένα συμβιβασμό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να μπορέσουμε εν συνεχεία να δεχθούμε μια οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων, επαναλαμβάνω σε περίπτωση όμως που καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Αυτή είναι η προϋπόθεση και έτσι πιστεύω μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο στο θέμα αυτό των ε, δικαιωμάτων των μετόχων, ταυτόχρονα δε να σεβαστούμε πλήρως ε, και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις εκθέσεις αναχώρα. Έρχομαι τώρα στα ψηφιακά. Ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές συμβάσει κτλ. Είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την οδηγία για τις επιγραμμικές πωλήσει. Θεωρούμε πως πρόκειται για ένα γενικό νομοθέτημα το οποίο έχει άμεση σχέση με την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, πιστεύω ότι οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Ήδη θα έχουμε, φαντάζομαι, μέσα στο καλοκαίρι τα αποτελέσματα της άσκησης REFIT. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς τις συζητήσεις μας τον Σεπτέμβρη πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια για να συνεχίσουμε πρέπει να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών. Κάτι που δεν θα συμβεί πριν το Σεπτέμβριο. Εξού και μιλώ για το Σεπτέμβριο ως ημερομηνία έναρξη αυτού του διαλόγου. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας, έτσι δεν είναι. Θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Προσβλέπω στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με εσά. Ίσως για το Βεξέλης 2 να πω ότι για μας είναι προτεραιότητα. Η Κομισιόν θέλει να ξεκινήσει συζητήσεις, είναι μια καλή προσέγγιση αυτή. Θέλουμε και εμείς να γίνει ένας διάλογος σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων και πιστεύουμε πως η Σλοβακία μπορεί να είναι ένας πολύ επικοδομητικός συνομιλητής. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις σας και τώρα το λόγιο ο κύριος Σέτσικ. Ο κύριος Κέστνερ έκανε μια ερώτηση για τον κανονισμό περί Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν εγκριθεί. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι είναι ώρα να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να γίνει εντό του φθινοπόρου. Εμείς θέλουμε να προετοιμάσουμε τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των τριμερών διαλόγων, κατά τρόπο ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί της Σλοβακικής Προεδρίας. Αυτό, αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημά σας. Το δεύτερο αφορούσε ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Η Κομισιόν δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων στις δημιουργικές βιομηχανίες. Είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Το 2014 ε, έγινε δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημιουργού, είναι σημαντικά και πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της προστασίας ε, των δικαιωμάτων των κατόχων ε, αυτών των δικαιωμάτων και των χρηστών. Θέλουμε ένα ισορροπημένο σύστημα. Θέλουμε δίκαιες απολαβές για τους δημιουργούς. Ε, θέλουμε δίκαιους όρους και συνθήκες και για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν είδη τα οποία είναι αντικείμενο προστασίας, προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα. Αναμένουμε το Σεπτέμβριο μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα ζητήματα. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε να επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα θέματα σε επίπεδο των ομάδων εμπειρογνωμόνων, τον οποίο και θα προεδρεύσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τα μέλη. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Οπότε να ευχαριστήσω εκ μέρου της επιτροπή μα και τους δύο διακεκριμένου καλεσμένους μας, την Υπουργό Δικαιοσύνη Λουτσία Ζητνιάσκα και τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιβάν Σετσίκ, που βρέθηκαν μαζί μας εδώ σήμερα και αναμένουμε να δούμε τα καλά αποτελέσματα της Προεδρίας σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας για λιγάκι να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 4 όπου θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτρόπο. 10 λεπτά λοιπόν διάλειμμα. Ευχαριστώ.

Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 26 της ημερησίας διάταξης. Να καλωσορίσω θα ήθελα την Επιτρόπο κυρία Μαρία Νετάσεν, Επίτροπο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα σε σχέση με αυτή η ανταλλαγή απόψεων σχετίζεται με τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας στο πλαίσιο της πρότασης για την απόσπαση εργαζομένων. Όπως ενημερώθηκα, η Επίτροπος υπήρξε μέλος της παρούσας Επιτροπής, οπότε διπλός ο λόγος για, για τον οποίο την καλωσορίζουμε μεταξύ μας. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω με εσάς ε, τη διαδικασία ελέγχου επικουρικότητα που έχει κινηθεί όπω γνωρίζετε στο πλαίσιο τη πρόταση μα για στοχευμένη τροπολογία τη πρόταση ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Η αρχική πρόταση συντάχθηκε πριν από 20 χρόνια για την απόσπαση των εργαζομένων. Στο μεταξύ οι συνθήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξελιχθεί και οι διαφορέ εντό τη Ευρωπαϊκής μα οικογένεια ε, έχουν διευρυνθεί. Για παράδειγμα, το 1996 η αναλογία, η αναλογία μεταξύ της ε, ελάχιστης και της μέγιστης ε, ε, αμοιβή ήταν ένα προς 3 και το 2016 είναι 1 προς 10. Η ανάλυση δείχνει ότι με αυτή τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των αμοιβών μεταξύ των κρατών μελών, οι κανόνες του 1996 για την απόσπαση των εργαζομένων οδηγούν ορισμένες φορές σε αθέμητα αποτελέσματα σε πίεση προς τα κάτω αντί για σύγκληση, σε έλλειψη δικαιοσύνης αντί για ίση αμοιβή. Και αυτό υπονομεύει την κατάσταση των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά. Για να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι μας να υποστηρίζουν την εσωτερική αγορά, όχι μόνο για τα αγαθά, αλλά και για τις υπηρεσίες, χρειαζόμαστε κανόνες σαφείς, δίκαιους και που να εφαρμόζονται στην πράξη. Κατά την άποψή μου, τέτοιοι κανόνε πρέπει να θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει λάβει η Κομισιόν αιτιολογημένε γνωμοδοτήσει από τα κοινοβούλια 11 κρατών μελών που εκφράζουν αμφιβολίε κατά πόσο η πρόταση τη Κομισιόν συμμορφώνεται με την αρχή τη επικουρικότητα. Σα διαβεβαιώ ότι το σήμα αυτό, το μήνυμα αυτό, εγώ το παίρνω πολύ στα σοβαρά. Έχουμε μελετήσει τι επιστολέ των διαφόρων κοινοβουλίων λεπτομερώ και Έχουμε ε, ξεκινήσει να συζητάμε τα ζητήματα αυτά με τα Εθνικά Κοινοβούλια και σε συναντήσεις που έγιναν στο Άμστερνταμ και στην Πρατισλάβα, στη συναντήση Κοζάκ. Ε, εγώ βρισκόμουν χθε στην Πρατισλάβα και είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ξέρετε, δεν είναι παρά η τρίτη φορά που η διαδικασία κίτρινης κάρτας ε, έχει ενεργοποιηθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για μια εξαιρετική ε, κατάσταση και εξετάσαμε όλα τα ζητήματα τα οποία έθιξαν τα ε, εθνικά κοινοβούλια. Μια από τις ε, πιο συνήθεις ενστάσεις ήταν ότι τα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της απόσπασης αντιμετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η απόσπαση εξορισμού είναι διασυνοριακή. Κατά συνέπεια, η ίδια δραστηριότητα έχει συνέπειες για τουλάχιστον δύο πλευρές ε, ενός σύνορου. Οι κανόνες λοιπόν για την απόσπαση αναγκαία δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ ατόμων σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Το να μην υπάρχουν κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο για την απόσπαση εργαζομένων οδηγεί σε σημαντική στρέβλωση της ελεύθερης διακίνησης ε, αγαθών και υπηρεσιών και ατόμων μεταξύ συνόρων. Και αυτό αναγνωρίστηκε από του συνομοθέτε το 1996 κατά την υιοθέτηση τη αρχική οδηγίας. Και πάλι το 2014 όταν συμφωνήθηκε η εφαρμοστική οδηγία, η εκτελεστική συγγνώμη οδηγία. Οπότε το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι κατά πόσο οι προτινόμενες αλλαγές είναι απαραίτητες και χρήσιμες ε, υπό το πρίσμα της επικουρικότητας. Εμείς θεωρούμε ότι οι στόχοι της πρότασης σίγουρα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Εάν τα κράτη-μέλη ε, δράσουν μόνο μερό σε εθνικό επίπεδο, για τις ε, αλλαγές που προτείνει το σχέδιο νομοθετικής πράξης θα οδηγηθούμε σε κατακαιρματισμό της ε, εσωτερικής αγοράς. Ε, βελτιωμένες συνθήκες ανταγωνισμού και επαρκής προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση είναι αδύνατο να διασφαλιστεί με δράση σε εθνικό επίπεδο μόνο. Άλλα σχόλια κύριε Πρόεδρε υπενήσονται ότι η πρόταση μπορεί να παρέμβει σε εθνικές αρμοδιότητες περί αμοιβή και βιομηχανικών σχέσεων. Αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η πρότασή μας δεν επεμβαίνει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων για τον ορισμό αμοιβών. Το μόνο που προτείνουμε είναι οι υποχρεωτικοί κανόνες που ε, ισχύουν για τους ντόπιου σε ένα κρατος μέλος και που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τι εθνικέ πρακτικέ στην αλληλόγω χώρο, ναι, ε, χώρα να ισχύουν επίση και για του αποσπασμένου εργαζομένου. Και ένα τελευταίο παράδειγμα σχολείων που έχουμε λάβει στι επιστολέ είναι ότι η πρότασή μα είναι πρόορη, διότι εμφανίστηκε πριν από την προθεσμία μεταφορά τη εκτελεστική οδηγία. Ε, προθεσμία που στο μεταξύ έχει παρέλθει από τις 18 Ιουνίου η εκτελεστική οδηγία υπήρξε ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Επίτευγμα στο οποίο συνέβαλε σημαντικά το παρόν κοινοβούλιο. Παρέχει στι εθνικέ αρχέ, νέα εργαλεία πολέμηση τη απάτη και των εταιριών γραμματοκιβωτίων. Ωστόσο, δεν ρυθμίζει το ζήτημα των ε, δίκαιων αμοιβών. Η πρότασή μας λοιπόν του Μαρτίου συμπληρώνει την εκτελεστική οδηγία, δεν τροποποιεί, ούτε παρεμβαίνει με αυτήν αξιότιμα μέλη, η Επιτροπή θα εξετάσει αυτό, τη διαδικασία ελέγχου της επικουρικότητας ε, όπως έχει προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα και θα αποφασίσει κατά πόσο θα αποσύρει, αν θα τροποποιήσει ή αν θα διατηρήσει την πρότασή μας. Να προσθέσω ότι η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τον πολιτικό διαλόγο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και πέραν αυτής της απόφασης. Οι συναδελφοί μου και εγώ ε, είχαμε πάνω από 300 συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια από την αρχή της εντολής μας και θα συνεχίσουμε την επαφή μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είμαι βέβαιη ότι το ζήτημα της δίκαιης εργασιακής κινητικότητας θα παραμείνει ε, από τις πρώτες προτεραιότητες του πολιτικού μας διαλόγου μέσα στα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες. Το πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή την ελεύθερη διακίνηση συνδυάζοντας την με δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού και επαρκή κοινωνική προστασία είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί επαρκώς δημοκρατικά σε ένα πλαίσιο όπου τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν τον λόγο τους μαζί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, το οποίο αποτελεί ένδειξη δημοκρατικής συζήτησης. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Είμαι πεπισμένη πολιτικά ότι η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη κινητικότητα και περισσότερε αποσπάσει εργαζομένων, όχι λιγότερε. Έτσι λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε τι συζητήσει μα για να δούμε πώ θα διασφαλίσουμε την ελεύθερη διακίνηση, συνδυάζοντά την με τη σωστή προστασία των εργαζομένων και ίσε συνθήκε ανταγωνισμού για τι επιχειρήσει. Εγώ προσβλέπω να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια όπου το καθένα από αυτά τα κοινοβουλία θα διδραματίσει το δικό του ρόλο σε αυτή τη δημοκρατική νομοθετική διαδικασία ευρωπαϊκού επίπεδου. Έχουμε ήδη κάνει πολύ καλέ συζητήσει για αυτό το θέμα με ευρωβουλευτέ ε, από όλε τι πολιτικέ οικογένειε, μαζί με του ε, σκιώδει συζητητέ, του συζητητέ και όπω γνωρίζετε το κοινοβούλιο αυτό μπορεί να υπολογίζει σε μένα. να Πάσα στιγμή μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα για να συζητήσουμε αυτό ή άλλα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγική σας παρουσίαση. Με την αδειά σα. Ε, θα έχουμε πολλές ερωτήσεις. Πρώτος ο κύριος Λοτόφσκι. Γεια σας, ε, καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, Υπάρχει ένα ερώτημα που σας έχω στείλει εδώ και καιρό, νομίζω τον Ιούνιο, και εσείς απαντήσατε το εξής. Η αλλαγή της οδηγίας εξερτάτε από τις ε, αρμοδιότητες των υπαλλήλων. Είναι δύσκολο ε, να ε, προβλεφθεί μια γενική ρύθμιση. Εκεί λοιπόν καθίσταται σαφές τι ακριβώς είναι το σχέδιο και τι ακριβώς ε, προβλέπετε εσείς. Λέτε πολύ σωστά ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, παρατηρήσεις για τα διάφορα κρατημέλη και αναλύετε εσείς αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν ελέγχθη όμως κατά πόσον εγκρίθηκαν ή όχι και αυτό θα αποφασιστεί μετά από μία εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, αυτές οι παρατηρήσεις θα εγκριθούν ή όχι. Και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση. Και έχω και άλλες τρεις ε, ερωτήσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιάζεται να προτείνει νέες ρυθμίσεις. Ε, πρόκειται για την ε, εφαρμογή μιας οδηγίας και πρόκειται και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο συζητάμε. Μετά ο στόχος αντιμετώπισης των παράνομων πρακτικών, αυτός είναι ε, πολύ καλός ε, και μία άλλη ερώτηση. Αυτές ε, οι αλλαγές οι διεθνείς μεταφορικές εταιρείες βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία στο προήμιο και μετά πρόκειται για τις ε, κοινωνικές διαβουλεύσεις και για την συγκέντρωση πληροφοριών σε σχέση με αυτή την πρόταση. Ε, και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς έγινε τελικά. Γιατί δεν, διαβα... δεν λαμβάνουν υπόψη αρκετές παρατηρήσεις από την κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ομολογώ ότι λυπούμε ιδιαίτερος. Συγγνώμη, μπορείτε κύριε Ποτόφσκι να κλείσετε το μικροφωνό σας. Κύριος Μπούντα, έλεγα λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος ε, μετά από τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου. Δεν στρέχουμε βέβαια εναντίον της Επιτρόπου, αλλά μιλώ γενικότερα για την Επιτροπή λίγο μετά το Brexit και φαίνεται ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πολλά πράγματα που έκριναν το αποτέλεσμα του υποψηφίσματος στη Βρετανία. Η Βρετανία μεταξύ άλλων επέλεξε να αποχωρήσει γιατί η Κομισιόν δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και πραγματικότητας στα κράτη-μέλη. Κυρία Επίτροπε, Έχετε παρατηρήσει από 11 κράτη-μέλη που λένε ότι η οδηγία παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Παρ' όλα αυτά όμως θέλετε να προχωρήσετε με την πρόταση αυτή. Έχετε μεν από πλευράς διαδικασίας τη δυνατότητα, αλλά δεν νομίζετε ότι τελικά εσείς παραβιάζετε τις αρχές της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη-μέλη μόνο μπορούν να, θεσπίζουν τους μισθούς ε, των εργαζομένων και αυτό σε συνάρτηση με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος. Πείτε μου λοιπόν, πώς θα διορθώσετε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν διαφορέ στου μισθού μεταξύ των χωρών Με Παραδείγματο χάρη, ο μέσο μισθό στην Ρουμανία είναι 400 ευρώ, ενώ στη Γερμανία είναι 2.000 ευρώ. Πώ μπορούμε να κάνουμε εναρμόνιση. Σας παρακαλώ σε εσά και όλους όσους είναι υπεύθυνοι, είναι αρμόδιοι να καταλάβετε. Να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια λύση, μια ενιαία λύση για όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι έχει κατάσταση. Και αυτό θα δημιουργηθεί με την οδηγία που δεν λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ε, του κάθε κράτους μέλους ή την ενιαία αγορά. Και δεν είναι η ίδια όλα τα κράτη-μέλη ως προς τις συνθήκες. Ευχαριστώ κύριε Μωρέν Σαχτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Τάισαν που ήρθε εδώ να μας ενημερώσει μετά τη συνάντηση της Μπρατισλάβα. Εγώ θέλω να σας πω ότι για το θέμα αυτό και είμαι πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω εργαστεί σε βάθος και για την ε, οδηγία, ε, την εφαρμοστική, σχετικά τον Απρίλιο του 2014. Βεβαίως δεν ήμουν μεταξύ αυτών οι οποίοι επιθυμούσαν η εν λόγω οδηγία του 1996 ε, να ξανασυζητηθεί, αλλά βλέποντας τη δική σας πρόταση, θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτα ισορροπημένη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να έχουν υπόψη. Δηλαδή, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής μας, σήμερα, μέσω της Ευρώπης, η κινητικότητα έχει γίνει ο κανόνας. Κινητικότητα των πολιτών, κινητικότητα των εργαζομένων είναι μία από τις αρχές στις οποίες εδράζεται η Ευρώπη μας. Και αυτό το οποίο εκτιμώ στην πρότασή σας είναι το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται από τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες προς τις δυτικές, αλλά και το ανάποδο. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία για τις διαφορετικές αυτές μετακινήσεις βλέπουμε ότι δεν είναι μονόδρομες ε, οι μετακινήσεις αυτές. Άρα νομίζω ότι νομίζω, ε, νομίζω λοιπόν ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Μια πρόταση ισορροπημένη λοιπόν η οποία αναγνωρίζει την αρχή της κινητικότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Αυτή η αρχή της κινητικότητας για μένα είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, κυρία Επιτροπή, διότι ακριβώς αυτή η κινητικότητα μα ε, μας δίνει τη δυνατότητα να αντισταθούμε στην ανεργία. Το επόμενο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι θεωρώ πως αν όλοι μπορούμε να εργαστούμε ισορροπημένα, με ανοιχτό πνεύμα και όλοι να συμφωνήσουμε, χωρίς εμπλοκές, με αυτή την οδηγία, την οποία θέλουμε να αναθεωρηθεί και να διορθωθεί μετά από 20 χρόνια. Εδώ θα έχουμε τα θεμέλια αυτή τη κοινωνική Ευρώπη. Σα άκουσα, αγαπητέ συνάδελφε, να λέτε ότι δεν καταλάβαμε τι μα είπαν οι Βρετανοί με τον Brexit. Εγώ σα απαντώ όχι, το αντίθετο. Όσο εδρεώνουμε την κοινωνική Ευρώπη, τόσο πιο ανθρώπινη απάντηση θα έχουμε να δώσουμε σε αυτούς που ψήφισαν υπέρ του Brexit. Μένα αυτό με ενδιαφέρει. Να μην ε, διαλυθεί η Ευρώπη από, ε, σε επίπεδο ανθρώπινο. Και εκεί εντάσσεται και εκεί δράσεται η δική μας δουλειά. Να βάλουμε τα θεμέλια για την κοινωνική Ευρώπη. Για να παραμείνουμε όλοι μαζί. Τέλος. Να προσθέσω κάτι ακόμη. Με το στόχο ακριβώς αυτό Πρέπει να συνεργαστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είδα ότι μου δείχνει το ρόλο σα. Λοιπόν, η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια είναι απολύτω απαραίτητη. Και ίσω είναι αυτό που δεν κάναμε μέχρι τώρα. Δεν ήταν αρκετά ανθρώπινη η Ευρώπη. Και ήταν πολύ μακριά από τα εθνικά κοινοβούλια. Βασιστείτε σε μένα για να εργαστούμε επικοδομητικά. Κυρία Χάταλα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο ότι η λύση είναι περισσότερο μια πιο έντονη εφαρμογή, εκτέλεση της οδηγίας, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι τόνισαν το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλά από τα κράτη-μέλη, όπως έχω υπολογίσει εγώ, τα 24 από τα 28, δεν έχουν κανονική κοινοβουλευτική εξέταση της δικής τους κυβέρνησης. Γι' αυτό τον λόγο δεν αντιμετωπίζουν ε, ε, στο πλαίσιο μιας τακτικής διαδικασίας ε, τέτοιες διαδικασίες όταν οι κυβέρνησεις ετοιμάζονται να υιοθετήσουν κάποια στάση για διάφορα νομοθετήματα στο Συμβούλιο. Ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί πιστεύω ότι θα βρούμε όλο και περισσότερες κίτρινες κάρτες και για καλούς λόγους Εκτός αν το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο αρχίσει να αποκτά ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά το να δίνει εντολή νομοθετική στην κυβέρνηση και πιστεύω ότι η κίτρινη κάρτα είναι το αντιστάθμισμα για την ανεπαρκή ε, επιρροή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν μόνο μία θέση στο Συμβούλιο. Ε, η κυρία Ουνισκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Το ζήτημα της απόσπασης εργαζομένων όπως βλέπουμε είναι ευαίσθητο, είναι υψηλής πολιτικής σπουδαιότητας για κάθε κρατός μέλος θα έλεγα. Ωστόσο, δεν είμαι βέβαιη για το πόσες από τις κίτρινες κάρτες που δίνονται αφορούν πραγματικά την επικουρικότητα. Γιατί ξέρετε, η επικουρικότητα μπορεί να θεωρηθεί από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όταν η δική μου χώρα, η Σουηδία, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας υποσχέθηκαν ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επηρέαζε το μοντέλο που διέπει τη δική μας αγορά εργασίας. Λόγω της ερμηνείας της σημερινής οδηγίας απόσπασης εργαζομένων, η Σουηδία δεν απολάβει την επικουρικότητα που τη είχαν υποσχεθεί. Τότε οι κοινωνικοί μα εταίροι ξέρουν καλύτερα από όλου ποιε κοινωνικέ συνθήκε απαιτούνται όταν ζει κανεί στη Σουηδία και θέλουμε οι κοινωνικοί μα εταίροι να μπορούν οι ίδιοι να καθορίσουν του κανόνες τη δική μα αγορά εργασία. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία για μα και πιστεύω επίση και ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να μπορούν να ανταγωνίζονται υποθεμητέ, ε, σωστέ συνθήκε ανταγωνισμού. Δεν είναι το θέμα η εναρμόνιση. Υπάρχει παρανόηση εδώ. Μιλάμε για ε, θεμητό ανταγωνισμό στην αγορά και ε, στην προκειμένη περίπτωση στην αγορά εργασία. Και αυτό δεν το έχουμε σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό η πρόταση τη Κομισιόν να προχωρήσει ώστε το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να τη συζητήσουν, να συζητήσουν τα πράγματα όπω έχουν σήμερα, ε, διότι δεν είναι βιώσιμα. Ευχαριστούμε, κύριε Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επιτροπέ. Ως εισηγητής ε, για την επικουρικότητα, για την Επιτροπή μας, εγώ ζήτησα την ακρόαση μέσα και χαίρομαι που η Επιτροπή μας και εσείς δεχτήκατε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι ε, πρώτα αναφέρθηκαν στην οδηγία του 96 και είναι μια, νομική μορφή που βρίσκεται σε κρίση. Αναφέρατε το ενεύλογη αιτία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, διαβίωση και ε, μισθού μεταξύ των κρατών μελών, μεγάλες διαφορές ε, κοινωνικών τελών και μια υπερβολική κινητικότητα εντό της Ένωσης οδηγεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Για να αναθεωρήσουμε λοιπόν αυτή την οδηγία, αναθεωρούμε αυτή την οδηγία διότι αντιληφθήκαμε το κοινωνικό dumping και είχε λάβει απαράδεκτα μεγάλες διαστάσεις. Τα πράγματα είναι σοβαρά, πρέπει να πω. Α δούμε το παράδειγμα τη Γαλλία, τη δική μου χώρα. Το 2015 είχαμε συν 25% αποσπασμένων εργαζομένων σε σχέση με το 2014. Με το προηγούμενο έτο είχαν αυξηθεί δηλαδή κατά 25% οι απασπασμένοι εργαζόμενοι είναι σχετικό όπως καταλαβαίνετε. Φτάσαμε λοιπόν σε μια πολιτική κρίση η οποία και γι' αυτό η συζήτησή μας σήμερα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση τις δυτικές χώρες που είναι υπέρ αυτής της αναθεώρησης μάλλον που την απαιτούν διότι ελπίζουν έτσι να περιορίσουν τον αριθμό των αποσπασμένων εργαζομένων και αφετέρου ε, τις ανατολικές χώρες ε, ε, ευχαριστώ κύριε Μαρασαρτιά αλλά ισχύει υποβάλλουν την κίτρινη κάρτα γιατί προσπαθούν να προστατεύσουν αυτή τη μορφή των αποσπασμένων εργαζομένων γιατί τους εξάγουν οπότε καταλαβαίνω απόλυτα τις απόψεις των μεν και των δε δεν θέλω να λαβω θέση βέβαια υπέρ η υπερ του αλλου Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίση. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει την ε, μεγάλη αγορά εργαζομένων, τη μεγάλη κινητικότητα εργαζομένων που ήθελε. Πρόκειται για μια τεράστια αποτυχία. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Εντάξει, ξέρετε, στην κίτρινη κάρτα τεχνικά υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία θα εξετάσετε. Η ιδέα αυτή της συλλογικής διαπραγμάτευσης, είναι ένα πολύ καλό ε, νομικό επιχείρημα. Ένα άλλο καλό επιχείρημα είναι ότι έχουμε περάσει από τον ελάχιστο μισθό που ήταν μια ε, ε, ευκολονόητη έννοια και συζητάμε πλέον περί ίσης αμοιβή για ίση εργασία σε ίδιο τόπο, κάτι που δημιουργεί προβλήματα. Είναι τεχνικά ενδιαφέροντα επιχειρημάτα, αλλά τίθεται το ζήτημα της επικουρικότητας. Ε, αλλά θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας και να σας ρωτήσω κατά πόσο συμφωνείτε. Μήπως δεν θεωρείτε κι εσείς ότι πέραν αυτό στις επιχειρηματολογίες έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Με το Brexit να είναι μόνο μια πτυχή όλο αυτού. Με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα αναδεικνύουμε το εξής πρόβλημα ότι δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη στην πραγματικότητα. Mr. Zwiefka. Κύριε Zwiefka. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję również pani komisarz za obecność. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για το ότι ήρθε και πάλι σε εμά. Ξανασυνδυόμαστε μετά από χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να αναφερθώ στο γεγονός ότι Τίτε το θέμα της αποζημίωσης. Όλα τα θέματα που τέθησαν από πλευράς περιεχομένου ε, δεν έχουν άμεση σχέση με αυτά που σας αφορούν. Όσον αφορά την επικουρικότητα θέλω να ρωτήσω ε, σχετικά με τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Μας ε, δώσατε συγκεκριμένες πληροφορίες ε, ε, θέλω να πω όμως ε, όλα αυτά που ακούσαμε με θλίβουν γιατί ήλπιζα ότι σήμερα θα ενημερωθούμε για το ποια θα είναι η αντίδραση της Επιτροπής. Και τώρα αυτό δεν έγινε και πρέπει να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Και υπάρχει άλλο ένα, ένα δεύτερο ερώτημα που αφορά και αυτό τις αρμοδιότητες της Νομικής Επιτροπής. Πρόκειται συγκεκριμένα για το εξής. Ε, πρόκειται για, τις, ε, για τα επικίνδυνα ε, προηγούμενα που αφορούν, που προέχουν από την, Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο άρθρο 2 εμφανίζεται κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται. Δηλαδή τροποποίηση των συμβάσεων αυτό ρυθμίζεται μέσα από τον κανισμό Ρώμη 1. Και αυτή η συμφωνία έχει άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή, οποτεδήποτε προσπαθεί κανείς να αλλάξει ορισμούς που περιλαμβάνονται στον κανονισμό Ρώμη 1, και αφορούν στον κανονισμό περί απόσπασης εργαζομένων, αυτά δεν είναι αποδεκτά. Παρακαλώ λοιπόν η Κομισιόν να μην το κάνει, να μην προσπαθεί να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Παρακαλώ λοιπόν να απευθυνθείτε στην νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λάβετε μία αδιαμφισβήτητη και ξεκάθαρη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αναφερθώ τόσο συγκεκριμένα σε νομικά θέματα όπως το έκανε ο Προλαλήσιας αλλά θα αναφερθώ σε κάποια ε, θέματα που έθιξε η κυρία Επίτροπος. Επισήμανε ότι λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν συνοριακά στοιχεία πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όσον αφορά στα προβλήματα αυτά, ε, πρόκειται για τους ελάχιστους μισθούς, για τις ε, εταιρείες ε, γραμματοκιβωτίου. Όλα αυτά βρίσκονται στην οδηγία και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Μιλήσατε για το γεγονός ότι οφείλουμε να ζητήσουμε μία αλληλέγγυα λύση. Σημαίνει αυτό το ίδιο Δηλαδή όταν μιλάμε για την ε, ελευθερία μετακίνησης ε, και παροχής των υπηρεσιών, τότε θα πρέπει να είναι ίδιο και το κόστος προσφοράς αυτών των υπηρεσιών. Κυρία Επίτροπε, ε, όσον αφορά τους μισθούς προτείνεται το εξής. Η Γαλλία έχει 32 επιδόματα επί του μισθού Δεν ξέρω αν τα έχετε ερευνήσει όλα αυτά, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι σε πάρα πολλά από αυτά τα επιδόματα υπάρχει επικάλυψη. Επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Και τι μπορεί να μας ε, προφυλάξει από το να υπάρχει αυτή η επικάλυψη των επιδομάτων, ας πούμε επιδόματα υγείας που επικαλύπτονται με επιδόματα διακοπών. Πολλά εξ αυτών όμως δεν καταβάλλονται από τους εργοδότες. Πώς μπορούμε λοιπόν ε, να προστατεύσουμε τους ε, εργαζόμενους και κάτι άλλο. Προτείνεται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να τεθούν επιτάπητο. Το σύστημα είναι αρκετά περίπλοκο. Ε, κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο, άλλες πάλι έχουν ε, τομεακές συμφωνίες, άλλες έχουν επιχειρησιακές συμφωνίες, επίπεδο επιχείρηση δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε διαφάνεια στον νομικ... στο τομέα της νομικής εφαρμογής και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία γιατί πιστεύω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προτάσεις οι οποίες μπορούν να ε, δημιουργήσουν δυσκολίες ε, στις εταιρείες αποστολής, μπορούν να οδηγήσουν σε κυρώσεις. Αν δούμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποσυρθεί κάποιες εταιρείε, μιλάμε για ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ. Ε, βλέπουμε λοιπόν πώς εφαρμόζεται ο προστατευτισμός. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήμουν ευγνώμων αν υπήρχε κάποια αναθεώρηση του όλου θέματος, κυρίως αν ε, δούμε λιγάκι τους αριθμούς και από εκεί διαπιστώνουμε τι είναι εκείνο που πραγματικά περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Πριν ε, λοιπόν δώσουμε το λόγο στην κυρία Επίτροπο, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήδη. Δηλαδή, στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων τίθεται το θέμα της επικουρικότητας. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, να τις ρωτήσετε στις συνεδριάσεις άλλων επιτροπών. Εδώ έχουμε να κάνουμε, εμάς μας ενδιαφέρει, η επικουρικότητα, το στοιχείο της επικουρικότητας που ενέχει αυτή η οδηγία. Η κυρία Ρέγνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ ευχαριστώ να κάνω αυτό που λέτε. Πράγματι πρόκειται για την επικουρικότητα. Όχι μόνο, αλλά κυρίως. Και γι' αυτό ε, θα κάνω και το εξή ερώτημα. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιφυλάξεις που εκφράζονται από ένα σημαντικό αριθμό κρατών μελών σχετικά με την επικουρικότητα, οι επιφυλάξεις αυτές να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Όμως, Όσον αφορά αυτές τις επιφυλάξεις, ακόμα και αν ε, υπάρχουν επιφυλάξεις από πλειοψηφία κρατών μελών, είναι σωστό να εκφράζονται επιχειρήματα που δεν ευστατούν, ακόμα και αν είναι πλειοψηφικό το αίτημα. Ας πάρουμε την οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα και εργάζονται σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι ε, κατά κύριο λόγο θέμα απόσπαση εργαζομένων και γι' αυτό πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως τα επιχειρήματα που εκφράζονται από κράτη-μέλη προφανώς και πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά κατά την άποψή μου ε, δεν υπάρχει κανένα θέμα που να είναι πιο διασυνοριακό και που να επιτρέπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να σκεφτούμε ότι εδώ πρόκειται για ε, συμφέροντα εργαζομένων στη χώρα Α, Β και Γ. Έτσι λοιπόν εξηγείται και το τι συμβαίνει, όπως είπε και ο κ. Μπούντα, στη Γερμανία ας πούμε μπορεί ο κατώτατος μισθέας σε ένα τομέα να είναι 2.000 ευρώ, αλλά σε άλλο τομέα 400 ευρώ. Και κατόπιν τούτου ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι ίδια μισθή για την ίδια δουλειά, στον ίδιο χώρο ε, και όχι να αναγκάζει κανείς ανθρώπους να κατεβαίνουν προς τα κάτω με τις μισθούς, να κάνουν dumping, αλλά να ανεβαίνουν προς τα πάνω, να ζητούν όλο και υψηλότερους μισθούς. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Τάισεν που λέει ότι η κοινή αγορά χρειάζεται κανόνες. Κυρίως όσον αφορά στην απόσπαση των εργαζομένων, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς διασυνοριακής ε, φύσης, άρα δηλαδή είναι απολύτως απαραίτητο όσον αφορά στην κοινή αγορά να τεθεί και το ερώτημα πώς συνδέονται όλα αυτά με κοινωνικούς κανόνες. Κατόπιν τούτου, από την εμπειρία μου, από τη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα από το δικό μου το κρατήδιο, τη Βόρειο Ιρανία έχουμε ένα νόμο ε, που λέει ότι πρέπει να είμαστε πιστοί στις συλλογικέ συμβάσεις. Σε εμά, στη Βόρεια Νέα Βεσφαλία, αυτός ο νόμος συνέβαλε στο να πιστούν θετικά οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή ότι πιστεύω αυτό είναι κάτι σημαντικό. Να πείσουμε τους ε, πολίτες για τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και να μην τους δίνουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη περιορίζεται μόνο και αυστηρά σε θέματα κοινή αγοράς. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Και εγώ θα ήθελα να περιστώ μόνο σε εκείνα τα ερωτήματα τα οποία αφορούν τη δική μας, τη νομική επιτροπή. Να στηρίξω το συνάλφο κύριο Τσέφκα που έπιξε το θέμα της επικουρικότητας και που ρώτησε μήπως μπορείτε λιγάκι να μας δώσετε έτσι μια γεύση του τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε. Την πρόταση θέλετε να τη διατηρήσετε, ε, σκέφτεστε τι μπορεί να αλλάξει ή τελικά πιστεύετε ότι καλύτερα την πρόταση αυτή να την αποσύρετε και να παρουσιάσετε κάτι τελείως καινούριο. Είναι σημαντικό για μένα να τα γνωρίζω αυτά και στηρίζει τον κύριο Σεύκα ε, που λέει ότι αν τελικά θέλουμε να αξιολογήσουμε διαφορετικά την επικουρικότητα να απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία ανεξάρτητα από το τι λέει η Κομισιόν ή οι τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις των κρατών μελών. Να κάνουμε εμείς τη δική μας τη δουλειά, ανεξάρτητη. Και έχω και μία ερώτηση κύριε Επίτροπε όσον αφορά την ε, ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ε, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου υπήρξε κυρία κίτρινη κάρτα ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων δεν είναι ικανοποιητική. Κυρίως οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη στο πλαίσιο της αξιολόγηση των επιπτώσεων. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε πιο συγκεκριμένα επ' αυτού. Κυρία Γλαμπάιωβα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Χαίρομαι που παίρνει πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό η Επιτροπή Γιούρη. Και έχετε δίκιο ότι υπάρχουν ε, πτυχέ που έχουν να κάνουν την απασχόληση, άλλα με το δίκαιο, νομικά θέματα, να μην τα αναμειγνύουμε όλα. Στην Επιτροπή Απασχόληση είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και μάλιστα με τη συνάδελφο Γιασλοβιέσκα οργανώσαμε και ένα σεμινάριο με εκπροσώπου Εθνικών Κοινοβουλίων, οι οποίοι ήρθαν και μα εξήγησαν τι δικέ του απόψει και μας παρουσίασαν τη συλλογιστική τους. Έχω δύο πολύ σύντομα ερωτήματα, διότι η Επίτροπος γνωρίζει πολύ καλά την άποψή μου και ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας αυτής. Όλοι μιλή, μιλάτε για την αρχή της επικουρικότητας. Υπάρχει όμως και μια άλλη πολύ βασική για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη. Αρχή που είναι η αρχή τη αναλογικότητα. Άρα, η ερώτηση προ την Επίτροπο είναι, η πρόταση αυτή είναι αναλογική σε σχέση με του στόχου που υποτίθεται ότι πρέπει να επιτύχει. Γιατί είναι και ένα σημαντικό επιχείρημα και αυτό. Δεύτερο ερώτημα, πιο πολιτικό αυτό. Δεν επισέρχομαι ούτε στι αρμοδιότητε Επιτροπή Απασχόληση, ούτε ε, στι αρμοδιότητε Επιτροπή Είναι πολιτικό το ερώτημα, σημαντικό για όλου μα. Σα ερωτώ, κυρία Επίτροπε, αν εσεί και το Σώμα των Επιτρόπων πήρατε σοβαρά ε, τα μηνύματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και η απάντηση δεν θα είναι αν θα προχωρήσετε ή όχι με την πρόταση. Το ερώτημά μου είναι από πολιτική πλευρά αν θα λάβετε υπόψη ε, τα μηνύματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά τα μηνύματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Τάισεν που είστε εδώ απόψε. Πολύ γρήγορα να σας πω, το 1996 Οπότε και τέθηκε σε ισχύ η πρώτη οδηγία για την αποσπάση των εργαζομένων που συζητούμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε 15 μέλη. 20 χρόνια μετά το 16 είμαστε 28. Προς το παρόν είμαστε ακόμη 28. Η μισθή το 96 ήταν ε, σε μια κλίμακα 1 έως 3 στην Ευρώπη των 15 και τώρα μιλάμε από 1 έως 12. Ε, περάσαμε από τη μια εποχή σε μια άλλη, από έναν αιώνα σε έναν άλλο ε, και στο πλαίσιο μιας καλύτερης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και της επαγγελματικής κινητικότητας, τι πιο λογικό ε, να σκεφτείτε τον εξοχρονισμό, την αναθεώρηση ε, της οδηγίας, ε, δηλαδή την παρουσίαση επικαιροποιημένων κανόνων και σε ό,τι αφορά την κλίμακα και σε ό,τι αφορά την οργάνωση, την εδαφική. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις σας περί αναθεώρησης της οδηγίας. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικές, πραγματιστικές και κινούνται ακριβώς με γνώμονα ε, την ανάγκη προσαρμογής ε, στις νέες ευρωπαϊκές πραγματικότητες. Δεν είμαι μέλος ε, του, της Νομικής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά και σέβομαι τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και τη σημασία τους και την ανάγκη να συμμετέχουν στις, στη λήψη αποφάσεων. Και πάντοτε παρακολουθώ με ενδιαφέρον και σεβασμό τι αποφασίζουν τα Εθνικά Κοινοβουλία. Και η συνάδελφος ε, Μωρέ και εδώ και σε άλλα ε, θέματα ακούσαμε επαρκώς τα Εθνικά Κοινοβουλία. Όμως θεωρώ ότι είναι προφανές όταν θέλουμε να ρυθμίσουμε την κινητικότητα των και γυναικών ε, εργαζομένων εντός ένωσης τη διασυνορική κινητικότητα κτλ. Τότε η αρμοδιότητα είναι ευρωπαϊκή για την οργάνωση και για την κυκλοφορία ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επικράτη. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστούμε πολύ. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Οπότε να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο να απαντήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και παρακαλώ επικεντρωθείτε όσο το δυνατόν στο ζήτημα της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για όλες αυτές τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, πήρα σημειώσει κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να δώσω απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έγιναν για το στοιχείο της επικουρικότητα. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να σα πω το εξή. Αυτή ήταν μια από τι πρώτε ερωτήσει. Κατά πόσο συνάδει με την εκτελεστική οδηγία που έπρεπε να μεταφερθεί μέχρι τις 18 Ιουνίου και η απάντησή μας είναι ναι. Είναι συμβατή, διότι η εκτελεστική οδηγία αφορά την εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης, ε, της κατάχρησης, ενώ η πρόταση που κάνουμε τώρα είναι μια πρόταση που ήρθε μετά την αναθεώρηση του ουσιώδους δικαίου των βασικών κανόνων της απόσπασης και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είχε έρθει η ώρα για μια αναθεώρηση, όχι πλήρη αναθεώρηση, στοχευμένη αναθεώρηση και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά λοιπόν την εφαρμογή ούτε τους σχετικούς κανόνες, αφορά, δεν αφορά να, αφορά να δώσουμε εργαλεία στα κρατημέλη να κάνουν καλύτερη εφαρμογή και να καταπολεμήσουν την απάτη αλλά και τους, εδώ αφορά περισσότερο τους ίδιους τους κανόνες. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα, η εκτελεστική οδηγία και αυτή εδώ η πρόταση, είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Τι άλλο έχουμε όσον αφορά την επικουρικότητα. Και τους μισθούς. Η πρόταση που κάνουμε συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας που έχει συμπεριληφθεί στη συνθήκη για τους λόγους που εξήγησα στην εισαγωγή μου. Να σας υπενθυμίσω οι, τις αντιδράσεις που βλέπουμε στις επιστολές των κοινοβουλίων που αφορούν την κίτρινη κάρτα. Σας έδωσα την απάντησή μου όσον αφορά τις αμοιβέ. Το τονίζω, η πρόταση αυτή δεν αφορά εναρμόνιση των αμοιβών και των μισθών στα κράτη-μέλη. Εναρμόνιση των μισθών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και σε πολλά κράτη-μέλη των κοινωνικών εταίρων. Αυτό διατυπώνεται σαφώς, θεσπίζεται στη συνθήκη την οποία εμείς τηρούμε. Δεν μπορεί η Κομισιόν ή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουν ε, πώς θα ορίσουν ε, μισθούς. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το μόνο που λέμε εμείς αυτή την πρόταση είναι ότι οι κανόνες περί μισθών, περί αμοιβών, οι κανόνες που εφαρμόζονται σε ε, εγχώριους εργαζομένους, εντόπους εργαζομένων, οι κανόνες που ισχύουν για αυτούς που έχουν θεσπιστεί ε, βάσει της νομοθεσίας ή με συλλογικέ συμβάσεις. Αυτοί οι υποχρεωτικοί κανόνες, λέμε, για τους ντόπιου εργαζομένους να είναι υποχρεωτικοί και για τους αποσπασμένους εργαζομένους που εργάζονται παράλληλα με τους ντόπιου στο ίδιο κρατός μέλος. Αυτό ζητάμε. Αυτό προσπαθούμε. Οπότε, όπως ακριβώς κάναμε και στην αρχική οδηγία του 96, ε, εκεί έλεγε ότι πρέπει να τηρείται ε, ο ελάχιστος μισθός. Όπως βλέπουμε, τα πράγματα δεν ισχύουν, δεν γίνονται έτσι σήμερα. Απλά εμεί λέμε ότι τα στοιχεία αμοιβή που είναι υποχρεωτικά για τους τοπικούς εργαζομένους να ισχύουν και για τους αποσπασμένους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αρχίζουμε να εναρμονίζουμε τους μισθούς. Αν πάτε και δείτε το κείμενο και το διαβάσετε προσεκτικά θα το καταλάβετε. Είναι κάτι διαφορετικό λοιπόν από αυτό. Να ευχαριστήσω την κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ήθελα να την ευχαριστήσω, αλλά μπορείτε να τη το μεταβάσετε, να το διαβάσετε. Να της διαβάσετε τις ευχαριστίες μου για τα πολύ θετικά τα σχόλια για την πρόταση μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι και εγώ έχω τη βούληση, όπως και όλοι οι συναδελφοί της Κομισιόν, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και καλό είναι που πρέπει το ίδιο και το Κοινοβούλιο με τις διάφορες επιτροπές. Ε, σκοπός μας είναι η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όποτε μας προσκαλούν πηγαίνουμε εκεί, εξηγούμε, πάντα είμαστε διατεθειμένοι να εξηγήσουμε τις προτάσεις μας είναι θέμα σεβασμού που υποχρεούμαστε να δείχνουμε ε, προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και έχουμε δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Για τις ε, παρατηρήσεις της κυρίας Άταλα, αυτό αφορά την εσωτερική οργάνωση, τον τρόπο με τον οποίο τα Εθνικά Κοινοβούλια συνεργάζονται με τα Υπουργεία τους. Δεν πρόκειται λοιπόν να σχολιάσω αυτό το θέμα να ευχαριστήσω και την κυρία Ουλφσκοκ για την υποστήριξη που εκφράσατε προς την πρότασή μας ε, λέγοντας ότι τηρεί τους κανόνες της επικουρικότητας. Το θέμα εδώ είναι να δημιουργηθούν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και επαρκής πρόσταση των αποσπασμένων εργαζομένων. Αυτοί ήταν οι δύο στόχοι που διακυβεύονταν όταν νομοθέτης το 1996 ή λίγο πριν αποφάσισε να κάνει κάτι για την απόσπαση και να λάβει σχετικές αποφάσει. Του ίδιου στόχου έχουμε και σήμερα. Μόνο που έχουν περάσει 20 χρόνια και θεωρούμε ότι απαιτείται μια στοχευμένη αναθεώρηση. Τι άλλο έχουμε. Uh, well, ε, Ah, euh, Κύριε Μπρετόν, ήθελα να πω ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της συνθήκης μας. Η πρόθεση λοιπόν των δυνατοτήτων αξιοποίησης αυτής της ελευθερίας αποτελεί σκοπό δικό μας, αποτελεί κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω και Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε ότι η εσωτερική αγορά δεν διέπεται από το νόμο της ζούγκλας. Η εσωτερική μας αγορά είναι μια αγορά οργανωμένη. Υπάρχουν κανόνες. Κανόνες για την κινητικότητα των προϊόντων, όπως και για την κινητικότητα των υπηρεσιών, για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και για την κινητικότητα των ατόμων, των προσώπων υπάρχουν κανόνες, υπάρχει οργάνωση. Γι' αυτό ε, μελετάμε κι εμείς ε, αυτή την πρόταση και την αναθεωρούμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς δίκαιους κανόνες οι οποίοι θα εφαρμοστούν. Αυτός είναι ο σκοπός της πρότασής μας. Κύριε Ζιασκά, ρωτήσατε ποια είναι η τελική μας αντίδραση, σε τελική ανάλυση όσον αφορά τις επιστολές που λάβαμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια των διαφορών χωρών. Όπως σας εξήγησα για την επικουρικότητα, πρώτα απ' όλα θα στείλουμε απαντήσεις σε όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια. Στο καθένα από αυτά θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που μας έχουν στείλει με τις επιστολές τους, είτε για θέματα επικουρικότητας, είτε για οτιδήποτε άλλο. Εμείς σίγουρα θα δώσουμε απαντήσεις ώστε να γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι, ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο της πρότασής μας. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση που πρέπει να λάβουμε από κοινού μαζί με όλους τους επιτρόπους ε, ε, στην Επιτροπή, εκεί η αντίδρασή μας θα βασιστεί στο μηχανισμό επικρουκότητας όπως προβλέπεται στις συνθήκες. Και εκεί θα αντιδράσουμε μόνο για το θέμα της επικουρικότητας, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε μια συνολική απάντηση για αυτό το θέμα του ελέγχου της επικουρικότητας. Εγώ ανέφερα τα τρία στοιχεία που βρίσκουμε να επαναλαμβάνονται σε αυτές τις επιστολές, τα οποία αναλύσαμε και είμαστε πεπισμένοι, συνεπώς, ότι έχουμε παραμείνει εντός των περιθωρίων ελιγμών που μας επιτρέπει η αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, ακούσαμε πολύ σαφώ τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν διάφορες γνώμες στα διάφορα κοινοβούλια. Ε, και ε, στα 11 κράτη-μέλη, τα κοινοβούλια των οποίων μας έγραψαν, ε, τονίζουν ότι δεν τους αρέσει η πρόταση για πολλούς λόγους που αφορούν το περιεχόμενό της. Από την άλλη λάβαμε και επιστολές από κυβερνήσεις, όπως και από κοινωνικούς εταίρους, άλλων κρατών μελών και κοινοβουλίων, που μας λένε ότι δεν θέλουν να ενεργοποιηθεί η κίτρινη κάρτα, διότι είναι πεπισμένοι ότι παίζουμε εντός των ε, περιθώριων της επικουρικότητας Οπότε βλέπουμε ότι κάποια κρατημέλη μάλιστα λένε ότι έχετε καθυστερήσει πολύ ή το παρατραβάτε. Άλλοι λένε τι κάνετε, είναι πολύ νωρί, ε, αυτό που προτείνετε δεν είναι αποδεκτό, το παρατραβάτε. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρότασή μα είναι μη ισορροπημένη, αλλά η συζήτηση είναι ανοιχτή. Όταν ξεκινήσουμε τη συζήτηση επί του περιεχομένου, η συζήτηση αυτή θα είναι εκτενής, δύσκολη, θα πάρει καιρό, αλλά θα χρειαστεί να συζητήσουμε μεταξύ μα, να ακούσουμε ένα τον άλλο για να δούμε που μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο, κάποιο συμβιβασμό επί όλων αυτών. Μια συμφωνία ε, στην οποία θα συνενεί η πλειοψηφία αφενός στο Συμβούλιο, αφετέρου στο Κοινοβούλιο. Έτσι νομοθετούμε στην Ευρώπη. Και έτσι πρέπει να πράξουμε με σαφή, διαφανή τρόπο. Εμείς τώρα λοιπόν θα μελετήσουμε τα στοιχεία της επικουρικότητας και αν αποφασίσουμε να συνεχίσουμε φυσικά θα γίνει εντελεχή συζήτηση εντός των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και με βέβαια θα παραμείνουμε σε επαφή με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης. Και φυσικά για το Σώμα των Επιτρόπων, εγώ θα προτείνω εκεί αυτά που πρότεινα το Μάρτιο. Διότι έχουμε κάνει έλεγχο επικουρικότητας και παλιότερα. Δεν είναι απλά έλεγχος ρουτίνας, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά. Ε, υποχρεούμεθα να το λάβουμε σοβαρά. Αποτελεί ακρογωνιαίο τη της ε, και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Ξέρετε, στην αρχή αυτής τη επιτροπή, ο κύριος Γιούνκερ είπε και ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι θα κάνουμε μεγάλα τα σημαντικά πράγματα και θα είμαστε μετριοπαθείς στα ε, μικρά πράγματα. Ο καθένας έχει την αρμοδιότητά του και θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το σωστό επίπεδο δράσης και για τους λόγους που ανέφερα στην εισαγωγή μου πιστεύω ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τι θα κάνουμε είναι το περιεχόμενο το οποίο θα ζητήσουμε περαιτέρω όταν θα μας δοθεί ευκαιρία. Τι άλλο ήθελα να πω για την επικουρικότητα. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς από εσάς. Πρέπει να πούμε σαφώς πιστεύω ότι η προστασία των εργαζομένων να έχουμε το ε, συνθήκε θεμητού ανταγωνισμού και την προστασία. Προστασία δεν σημαίνει προστατευτισμό. Πρέπει να είμαστε σαφοί. Εγώ ποτέ μου σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποστηρίξω τον προστατευτισμό. Εγώ μεγάλωσα μέσα στην εσωτερική αγορά. Σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και είμαι πεπισμένη για τα ωφέλη μια οργανωμένη ενιαία αγορά. Ο προστατευτισμό δεν έχει καμία θέση στη δική μα ενιαία αγορά. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ρέκνερ και Κώστερ που έκαναν ε, πολύ θετικά σχόλια και συμφωνούμε για το πώς χειριζόμαστε ε, και πώς προτείνουμε να ξεκινήσει μια συζήτηση. Επίσης ε, έκανε μια ερώτηση κυρία Λίμπερ για το κατά πόσο στην εκτίμηση αντικτύπου μας εξετάσαμε επίσης την περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ναι, σας καλούμε να διαβάσετε την εκτίμηση αντικτύπου και φυσικά όπως γνωρίζετε η μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη και βρίσκονται στο επίκεντρο των δικών μου πολιτικών. Εμεί πραγματοποιήσαμε την εκτίμηση αντικτύπου για να δούμε ποιε θα ήταν οι συνέπειε και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, τόσο εκεί όπου βρίσκονται, όσο και εκεί που φιλοξενούνται για να παράγουν υπηρεσίε. Τώρα, όσον αφορά την επικουρικότητα, να συμφωνώ, η νομική υπηρεσία μπορεί να ρίξει μια ματιά, είναι λογικό. Έχουμε κάνει αυτή την αξία και εντός της δικής μας δομικής υπηρεσίας και μετά έχουμε και την άλλη παρατήρηση. Ε, ξέρετε, έχουμε και το θέμα του Ρώμη 1. Ε, μετά από συμβουλές από τους νομικούς μας συμβούλους είδαμε ότι συμμορφώνεται με το Ρώμη 1 για το ποια νομοθεσία εφαρμόζεται, ποια χρονική στιγμή αλλά ξέρετε στο πλαίσιο του Ρώμη 1 όταν υπάρχει υποχρεωτική νομοθεσία η οποία παρέχει καλύτερη προστασία σε έναν εργαζόμενο, ο εργαζόμενος μπορεί να υπολογίζει σε αυτό. Οπότε αυτό ισχύει και σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις ε, για τα θέματα επικουρικότητας και λίγο παραπάνω. Ελπίζω να κατέστησα τα πράγματα πιο σαφή όσον αφορά την πρότασή μας και να σα εξήγησα επαρκώ του ε, στόχου και τι αιτίε που μα οδηγούν σε αυτή την αναθεώρηση, τη στοχευμένη αναθεώρηση. Ελπίζω ότι τα πράγματα είναι πιο σαφή και για τα μέλη εδώ τη Επιτροπή Δημοκρατικών Θεμάτων. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε και εμείς την Επίτροπο που ήρθε σήμερα κοντά μας και απάντησε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που σας υποβάλαμε και είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούμε στο μέλλον, ίσως όχι αυτό το θέμα, ενδεχομένως για κάποιο άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε μετά από το αίτημα του κυρίου Ζεύκα με το 11. Ε, ανταλλαγή απόψεων για... Ε, την αφαιρεγγιότητα, διαδικασίες αφαιρεγγιότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. Και όποιος θέλει ε, μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση του εκτός έτους. Κύριε ε, Ζεύκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και λυπούμε πολύ που έκανα αυτό το αίτημα, αλλά χαίρομαι που αποφασίσατε να με ακούσετε. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή της ε, περίοδου αυτής ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για έναν κανονισμό για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Ουσιαστικά, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα θα είναι συνέπεια της ε, έγκρισης των λόγου αυτού εγγράφου όλα όσα συμβαίνουν, συμβαίνουν σε επίπεδο κρατών μελών. Εγώ προσπαθώ να σας περιγράψω ουσιαστικά μια αμυγός τεχνική τροποποίηση. Δεν έχει δηλαδή νόημα να συζητήσουμε κάτι. Στην Πολωνία στο μεταξύ το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του ζητήματος και τη μεταφορά των σχετικών διατάξεων περιφερειακών στο εθνικό δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση στην Πολωνία. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες λοιπόν ε, αφαιρεγκαιότητα και υπάρχουν και συγκεκριμένοι επαγγελματίες ε, τους οποίους αφορά αυτή η αλλαγή και θα πρέπει στα παραρτήματα του κανονισμού να αντικατοπτρίζονται αυτές οι αλλαγές. Είναι δύο τα παραρτήματα το πρώτο περιλαμβάνει τον κατάλογο των διαδικασιών, το παράρτημα Α και υπάρχει και ένα δεύτερο, το παράρτημα Β, με ένα κατάλογο των διαχειριστών αυτών των διαδικασιών. Παραλαμβάνω, είναι το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης στην Πολωνία και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είπε ναι, δέχθηκε τις αλλαγές αυτές, ωστόσο, με βάση την ισχύουσα διαδικασία και επειδή η απόφαση πρέπει να είναι κοινή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε. Όπως είπα, είναι τεχνικό το ζήτημα επί της ουσίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω το εξής χρονοδιάγραμμα. 5 Σεπτεμβρίου αμέσως μετά το καλοκαίρι στην πρώτη μας συνεδρίαση να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο έκθεσης και ενδεχομένως να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Τεχνικό επαναλαμβάνω το θέμα. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών, δυστυχώς επειδή πρέπει να είναι έτοιμο το κείμενο πιο πριν και αν έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο φθινόπωρο τη εργασία μα. Δεν μπορεί λοιπόν η προθεσμία να είναι μεγάλη γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό και να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ του εγγράφου και των προτινόμενων αλλαγών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σα ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσει από τους ε, συναδέλφου. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο το λόγο. Είχαμε μια μονομερή ανταλλαγή απόψεων. <laughs> Ευχαριστώ τον κύριο Τσβέφκα και περνάμε στο επόμενο, στο σημείο 10. Γυρίζουμε πίσω. Ερμηνεία και υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας. Είμαι η από κοινού με τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα σας αναφέρω συντομία τι ε, γίνει στις δύο συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για την ερμηνεία και υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας. Συγκεκριμένα 7 Ιουνίου η ομάδα εργασίας εστίασε σε τρία βασικά ζητήματα. Τα εξής πιθανές ω κανόνες στο εσωτερικό οργανισμό του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, πρόγραμμα, προγραμματισμό Τρίτον, επαλήθευση νομικών βάσεων. Αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν παρουσία του κυρίου Μπούζεκ και του κυρίου Βίλαντ που προεδρεύει τη Ομάδα εργασίας Επιτροπής για τον εσωτερικό κανονισμό. Ο κύριος Μπούζεκ ανέφερε τις βασικές προκλήσεις ε, που δημιουργεί η Διοργανική Συμφωνία στον τομέα του προγραμματισμού. Ο κύριος Μπούζεκ ανέφερε ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να έχουν διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και την επιτάχυνση των νομοθετικών εργασιών. και θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν τα χρονοδιαγράμματά τους άλλοι φορείς, άλλα θεσμικά όργανα. Σε ό,τι αφορά τις νομικές βάσεις, ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων ή διακανονισμών για την Διοργανική Συμφωνία ή αρμοδιότητες επιτροπής μας θα πρέπει να διατηρηθούν απολύτως. Συμφώνησε ο κ. Σκορμπέτ από αυτού. Είπε ότι αυτό συγκλίνει και με τις δικές του Προτάσει τροπολογιών για τον ιστορικό κανονισμό. Διευκρίνησε επίσης ότι όταν υπάρχει ανταλλαγή απόψε με άλλα θεσμικά όργανα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί το εν λόγω καθήκον να το αναθέτει στον πρόεδρο της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι και αρμόδια Επιτροπή για την Επαλήθευση των Νομικών Βάσεων. Η ομάδα εργασία συνεδρίασε και στις 4 Ιουλίου. Εκεί υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με τον Έλμαρ Μπροκ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και με τον Μπεντ Λάγκε, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Θέμα ήταν βελτιωμένες πρακτικές ρυθμίσεις για την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τη σύννεψη διεθνών συμφωνιών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 40 της Νέας Διοργανικής Συμφωνίας. Ο κύριος Λάγκη λέει ότι οι διαπραγματευτές θα πρέπει να έχουν επαφή με Λίμπετραν, Πέσ ΕΝΒΙ, ΑΦΚΟ, Γιούρι. όπως και με τη διάσκεψη των πρώτων των Επιτροπών. Και θα πρέπει να αναφέρουν στην διάσκεψη των Προέδρων. Πρώτη συνάντηση με τις Αλόγω Επιτροπές έγινε στις 22 Ιουνίου και συμμετείχα και εγώ. Αναφέρθηκε συντομία στα σημαντικότερα προβλήματα και δυσκολίες. Πρέπει να υπάρχει έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες και στα έγγραφα και να μην θεωρούνται διαβαθμισμένα ε, κάποια έγγραφα αχρίαστα αν αλλάξει νομική βάση. Ο κύριος Λάγκε αναφέρει επίσης ε, την πρόσφατη απόφαση ε, για την Τανζανία. Ευνοϊκή για το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πληροφόρησης και είπε ο κύριος Λάγκε ότι ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία τη Σλοβακική Προεδρίας. Μετά πήρε το λόγο ο κύριος Μπρόκ, ο οποίο πρόσθεσε ότι θα γίνουν συναντήσεις με τις επιτροπές ή μάλλον θα γίνονται ε, συναντήσει με τι επιτροπέ πριν και μετά κάθε διαπραγματευτικό κύκλο. Και οι πρόεδροι των επιτροπών ενδεχομένω θα προσκαλούνται να ε, συμμετάσχουν εφόσον ε, συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα τις επιτροπές και είπε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στην στήριξη των επιτροπών Γιούρι, Αύκο και βέβαια και των άλλων επιτροπών. Έπειτα, η ομάδα εργασία συζήτησε την ομολογία του δικαστηρίου. Το πρόβλημα για τη χρήση μυστικών εφουσών ανάγνωσης, TTIP, διαμεσολαβήτρια και η αρχή need to know και οι μεικτές συμφωνίες ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε. Τώρα, το κατά πόσο συμφωνία είναι μεικτή ή όχι, Θεωρώ ότι είναι διαπραγμάτευτο το θέμα ο κύριο Μπρόκ και δεν θα πρέπει να μπει στο θεματολόγιο των διαπραγματεύσεων για το πρωτογενέ δίκαιο κτλ. Ε, Επίση, εγώ ανέφερα ότι υπάρχει ίσως ε, παράπλευρη απώλεια με τη διαφάνεια, δηλαδή ότι μπορεί να αποκαλύπτουμε κάποιες κόκκινες γραμμές ε, στις διαπραγματεύσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δύο τελευταίων συνεδριάσεων της ομάδος εργασίας μας. Η κυρία λέμε πως θέλει κάτι να προσθέσει. Ε, well. Κοιτάξτε, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή στην οποία αναφερθήκατε και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτά τα οποία ορίστηκαν ως δικαίωμα του Κοινοβουλίου ε, για την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν σε διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες, αυτό το δικαίωμα ε, δεν είχε καταρχήν προβλεφθεί. Και αυτή η ιδέα του να υπάρχει ένας χώρος, μια αίθουσα για να μπορεί κανείς να διαβάσει έγγραφα ήταν για ευαίσθητα έγγραφα εξωτερικής πολιτικής του τρίτου πυλώνα ε, τότε που ε, τα θέματα αυτά δεν ενετάσοντο μέσα στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν το δικαίωμα του να είναι κανείς πλήρως και έγκαιρα ενημερωμένος. Άρα δηλαδή το Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκε γιατί νομίζω ότι έχει προάγει την ε, πρόσβαση, τη δυνατότητα πρόσβασης του Κοινοβουλίου σε έγγραφα στο βαθμό που μπορούσε και το ίδιο είχε κάνει και η Επίτροπος κυρία ε, Μάλμα. Και τώρα ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, παραδείγματο χάρη στι διαπραγματεύσει για το TTIP, έχουν βάλει ένα όριο για το πόσα και ποια έγγραφα μπορούμε να μελετάμε. Άρα δηλαδή εδώ πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που έχει σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες. Και εμεί ευχαριστούμε. Άλλος παρακαλώ, από ό,τι βλέπω όχι, άρα κλείνει και αυτό το θέμα και πάμε στο υπαριθμόν 29. Εδώ πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ε, συμβάσεις ε, για την επιγραμμική ε, και εξαποστάσεως πώληση αγαθών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας είχα υποσχεθεί ότι αυτή η νομοθετική άσκηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να δείξω λιγάκι υπομονή καθώς θα προσπαθώ να εξηγήσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δύο νομοθετικές προτάσεις στις 9 Σεπτεμβρίου που αφορούν στην ψηφιακή κοινή αγορά. Η μία αφορά στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου και η άλλη, με αυτήν ασχολούμαστε τώρα εδώ, πρόκειται για την επιγραμμική και εξαποστάσεως πώληση ενσωματώσεως σώμα των αγαθών, ας πούμε παπούτσια, ηλεκτρικές ε, συσκευές, οτιδήποτε. Οι δύο προτάσεις είναι πολύ στενά συνδεμένες μεταξύ τους και στο επίκεντρο της των συζητήσεων ανάμεσα στους συγητές και τους σκιώδης συγητές των δύο προτάσεων υπάρχει αυτή η αλληλένδετη σχέση των δύο προτάσεων και κατ' ουσίαν γι' αυτό ζήτησα από τη Σλοβάκα Υπουργό να μας πει κατά πόσο προτίθεται να επιταχύνει λιγάκι στο Συμβούλιο τις ε, συζητήσεις σχετικά με την πρόταση περί ενσώματων αγατών. Η δουλειά για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, είναι ήδη πολύ προχωρημένη και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την διασύνδεση. Ο κύριος Φως ε, που είναι ο ε, εισηγητής ε, αυτού του ψηφιακού περιεχομένου τα γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά. Ε, μέχρι τώρα η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή ανάμεσα στους συναδέλφους και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ έτσι λοιπόν το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι το εξής. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας ε, των ε, καταναλωτών σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η Κομισιόν προτείνει να εξετάσουμε ξεχωριστά το ψηφιακό περιεχόμενο και τα ενσώματα αγατά και ο διαχωρισμός ε, είναι λογικός όταν είναι σαφές το περιεχόμενο, αλλά δεν είναι πάντα, δεν ισχύει πάντα αυτό και η πολυπλοκότητα δεν επιτρέπει να διαχωρίζει κανείς ε, τα ε, διάφορα νομικά καθεστώτα. Ας πούμε, σαν παράδειγμα, το smartphone είναι και αυτό ένα τηλέφωνο, αλλά κυρίως αποτελείται από λογισμικό που πρέπει κανείς να το ε, ενημερώνει συχνά. Ή ένα έξυπνο ψυγείο, ε, όταν σταματήσει να λειτουργεί, ίσως αυτό να οφείλεται και πάλι στο ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό του. Η δυσκολία λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη και θα προκύψει περισσότερο στο μέλλον ε, σε σχέση με το διαδίκτυο και τη ρομποτική. Αυτά αποκαλούνται και κυβερνοφυσικά συστήματα, cyber physical, εμείς λοιπόν ε, στην Επιτροπή Τζούρι και προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε να βρούμε την εμβέλεια αυτών των δύο προτάσεων. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα δύο καθεστώτα στο βαθμό του δυνατού έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην αντιμετωπίζουν σύγχυση ε, και να έχουν νομική ασφάλεια. Καθοριστικό αυτό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην περιορίσουμε το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στην Ευρώπη. Πρέπει να παραμείνει υψηλό το επίπεδο αυτό, γιατί για σκεφτείτε τι θα συμβεί όπως συνέβη με την προηγούμενη πρόταση που δεν θυμάμαι ακριβώς ε, πώς τη λέγανε ε, η οδηγία περί κοινών ε, πωλήσεων πρόκειται για την εναρμόνιση. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε ε, έξυπνες λύσεις ε, τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ήδη ε, ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και στις πωλήσει και αυτό πρέπει να θεωρείται ως ένα κεκτημένο. Όσον αφορά λοιπόν τις νομικές προτάσεις, αυτές είναι πάρα και θα θυμάστε εδώ ένα παράδειγμα του τι δεν πήγε καλά. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, πολλές και διαφορετικές προτάσεις από την Επιτροπή που θίγουν θέματα που δεν έχουν μέχρι τώρα εξεταστεί από το δίκαιο των συμβάσεων. Ψηφιακά ή μη ψηφιακό περιεχόμενο, ε, προστασία δεδομένων. Αυτό μέχρι τώρα το ε, διασφαλίζει είναι ψηφιακο περιεχομενο προστασια περί προσωπικών δεδομένων μιλάμε για την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες χωρί να πληρώνουν με χρήμα. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε μια σωστή εναρμόνιση. Παραδείγματο χάρη, σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει περίοδο νομική εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζουν. Όμω, ε, τα ωφέλη για τους καταναλωτές ε, θα πρέπει να είναι πάνω από δύο χρόνια αν και η διάρκεια ε, ζωής ε, των προϊόντων θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που πολλά εξ αυτών έχουν διάρκεια ζωής πάνω από δύο χρόνια οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η διάρκεια ζωής τους θα είναι πολύ μεγάλη δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τις νόμιμες προσδοκίες των καταναλωτών άρα κατέληξα ε, στο ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι την ε, περίοδο της ε, νομικής εγγύησης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με βάση την οδηγία Equal Design εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα ιδέα. Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό δίκο, δίκαιο, αλλά και με μια νέα ιδέα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ε, αντεκτικότητα και την διάρκεια ζωή. Δύο βασικά στοιχεία αυτά να περιλαμβάνονται μέσα στη σύμβαση. Και αυτό έχει σχέση βέβαια και με την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει με την βιώσιμη κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ σύντομα να σας αναφέρω και το χρονοδιάγραμμα για όλη αυτή την ε, εργασία. Επειδή συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους μας που είναι αρμόδιοι για το ψηφιακό περιεχόμενο, έχουμε προσαρμόσει λιγάκι το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσουμε από κοινού. Και θα σας παρουσιάσω ε, σχέδιο έκθεσης ε, το Σεπτέμβρη και έτσι λοιπόν η προθεσμία για ε, τροπολογίες είναι 26 Οκτωβρίου. Οι τροπολογίες θα εξεταστούν από τις 28 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία για το σχέδιο της γνωμοδότησης στην Τζούρι θα λάβει χώρα ε, στις 17 Ιανουαρίου και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια. Πάντως με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις σας και επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία με τον κύριο Φόρσε που είναι εισηγητής ε, του ε, ψηφιακού περιεχομένου, της σχετικής οδηγίας δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Χάταλα για την παρουσίασή της. Λίγα λόγια κύριε Πρόεδρε, κοινή μας φιλοδοξία είναι να προσφέρουμε ένα πλαίσιο το οποίο ταυτόχρονα θα είναι ασφαλές και απλουστευμένο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και που θα προσφέρει προστασία στους καταναλωτές μας ώστε να αξιοποιήσουμε σε όλη τους την έκταση τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση των ανταλλαγών, των συναλλαγών ε, εντείνοντάς και αναπτύσσοντάς η κυρία Χατάλα παρουσίασε πολύ σωστά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο προτάσεις ε, παράλληλες ε, που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διακρίνω ευνοϊκές εξελίξεις για τους καταναλωτές μεταξύ των οποίων βρίσκουμε κυρίως την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης όπως βλέπουμε στο σχέδιο είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, όσον αφορά τα διάφορα διακυβεύματα που αναφέρθηκαν, θα δούμε ότι εξετάζονται με μεγάλη προσοχή και σε βάθος, όπως είπε και η κυρία Συγήτρια. Βλέπουμε ότι θέλουμε την απλούστευση της εσωτερικής αγοράς, την ευελιξία μαζί με την εναρμόνιση καθώς και τη βούληση να διατηρήσουμε στα κράτη-μέλη διατάξεις ε, υψηλού επίπεδου προστασίας για τους καταναλωτές. Αυτά θα αποτελούν τους στόχους μας. Υποστηρίζουμε τους συνεισηγητές ΙΜΚΟ ε, και Τζούρι ε, και την εργασία του εισηγητή ΙΜΚΟ για την οδηγία πωλήσεων online Όσοι δηλαδή εργάζονται και για τα δύο κείμενα και στις δύο επιτροπές θα πρέπει να έχουν την όσο το δυνατό πιο συνεκτική προσέγγιση και για τις δύο προτάσεις κειμένου και να δουν πώς θα μπορούσαν να προσαρμόσουν, να κάνουν να συγκλίνουν τα διαφορετικά νομικά πλαίσια που ισχύουν στο πλαίσιο των καταναλωτών σε σχέση με ό,τι συμβαίνει ε, εκτός διαδικτύου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να προσέχουμε τυχόν σύγχυση μεταξύ των δύο κειμένων, να ξεκαθαρίσουμε ε, ε, και να διαχωρίσουμε σαφώς ε, τα πεδία εφαρμογή των δύο προτάσεων, να βρούμε τα κοινά σημεία, να βρούμε τις συγκλήσεις, να επιλύσουμε τη σημεία σύγχυσης. Έχουμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο θα μας δώσει χρόνο σκέψης και σύνταξης των ενδεχόμενων τροπολογιών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, κύριο Τζαμπάσκι. Благодаря, господин Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Χάουταλα. Χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να πω την άποψή μου για αυτό το πολύ σημαντικό ε, θέμα. Επειδή σκοπεύουμε να εναρμονίσουμε τις συμβάσεις online, πρέπει να προβούμε σε, σε βάθος ανάλυση του θέματος. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να προειδοποιήσω όλους μας ε, να μην δράσουμε υπερβολικά γρήγορα και απερίσκεπτα. Το Ρίφιτ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα αναμένονται το φθινόπωρο. Και ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε απόφαση που θα αφορά την ενιαία αγορά πρέπει να αναλυθεί και από την άψη του Refit. Επίσης θα πρέπει να δούμε και κάποιες πτυχές των πωλήσεων ε, προϊόντων στο διαδίκτυο. Αν βιαστούμε υπερβολικά τώρα και δεν περιμένουμε το refit, θα δημιουργηθεί ακόμη περισσότερη σύγχυση. Όσον αφορά τις ε, διαδικτυακές πωλήσει. Βλέπω πολλές λεπτομέρειες εδώ και θέλω να πω ότι η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπέρ αυτών των μέσων υπεράσπισης των καταναλωτών. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τους ορισμούς και να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τους ορισμούς αυτούς προς όφελος των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ο στόχος μας ανά πάσα στιγμή. Και σε όλες τις περιπτώσεις οι καταναλωτές πρέπει να κερδίζουν σε, από αυτές τις συμβάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος του κειμένου φυσικά και είναι αξιέπαινος. Ποιος είναι κατά ε, της προστασίας των καταναλωτών στις διαδικτυακές δεσμευτικές πωλήσει. Όμως, όταν διαβάζουμε την πρόταση οδηγίας ε, αμφιβάλλουμε λίγο παραπάνω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω των συνθήκων ουσιαστικά θα γίνω εκπρόσωπος ε, φερέφωνο της γνώμης ε, της Ιταλικής της ε, Γαλλικής Γερουσίας. Στην πρώτη Οδηγία. έχουμε το άρθρο 3, επίπεδο εναρμόνισης, που πιέζει πραγματικά προς μια πολύ μεγάλη υπερβολική εναρμόνιση. Απαγορεύει τα κράτη στο εθνικό δίκαιο να εισαγάγουν διατάξεις που αποκλίνουν από αυτές τις οδηγίες μεταξύ αυτών πιο αυστηρές ή πιο ευέλικτες διατάξεις. Δηλαδή, τι λέμε με άλλα λόγια, ασφυξία ε, δημιουργούμε, ε, στραγγαλίζουμε. Ε, τι λέει λοιπόν η πιο ευελικτε διαταξεις δηλαδη τι λεμε με πολύ σωστά. Αν δεν τηρήσουμε το άρθρο 3 έχει, εγγυήσεις που αυτή τη στιγμή παρέχει το γαλλικό, ο γαλλικός αστικός κώδικας ε, πάβουν πλέον να ισχύουν. Άρα, ναι, μεν θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, αλλά ακριβώς για να τους προστατεύσουμε, ε, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Όχι να μειώσουμε την προστασία τους, στο επίπεδο σας που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Άρα προσοχή στο άρθρο 3. Ευχαριστώ. Κύριος Φως. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Την εισηγήτρια. Έχουμε εργαστεί πάνω στο θέμα και έχουμε δει τη διαφορά μεταξύ των ψηφιακών και των ενσώματων αγαθών. Κάποιες φορές, όπως είπε και η συγγήτρια, τα πράγματα είναι λεπτά και έχουμε όλο και περισσότερα ενσώματα αγαθά που σχετίζονται με λογισμικά ή άλλες λειτουργίες, άρα η διάκριση καθίσταται όλο και πιο δύσκολη. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να εισαγάγουμε μια αρκετά λογική διάκριση. Σήμερα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Πού θα επιτρέπει αυτή τη διάκριση. Θέλουμε επίση να έχουμε μια γενική προσέγγιση που θα ενσωματώνει και συναφεί ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό θεματολόγιο. Έχουμε τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων, την οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενδεχομένως και άλλα. Άλλα θέματα. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια προσέγγιση των διαφορετικών θέσεων. Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις καλό είναι να βρούμε ένα κοινό έδαφος συνεννόησης. Και επειδή μιλάμε και για το επιγραμμικό περιεχόμενο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είναι στο δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση, να μην πω πλήρη ε, η εναρμόνιση, διότι ε, όλο και περισσότερη διασύνδεση έχουμε. Καλό είναι λοιπόν να βρούμε μια κοινή λύση για να αποφύγουμε χάσματα. Υπάρχει επίσης η εναρμόνιση των νομοθεσιών, διακρίσεις μεταξύ ψηφιακού, ενσώματου κτλ. Τα είπα και τα ξανά είπα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ λοιπόν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αρκετά μεγάλη εναρμόνιση. για να μην έχουμε τελείως διαφορετικές νομικές οδούς, να μην έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις, άλλα να ισχύουν για τις διαδικτυακές πωλήσει, άλλα για τα δικαιώματα, προστασία, καταναλωτή κτλ. Και να μην έχουμε ένα κατακαιρματισμό. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ ο κύριος Ράντιεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αποφεύγουν τις διαδικτυακές αγορές διότι αμφιβάλλουν κατά πόσο προστατεύονται τα δικαιώματά τους και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Έτσι διστάζουν να πραγματοποιήσουν ε, διασυνοριακές αγορές. φοβούνται τα προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που διαμαρτυρηθούν ή σε περίπτωση μη παράδοση των αγορών του. Κατά συνέπεια το νέο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσει που συνεπάγεται αυτό ο νέος δυναμικός τομέας, μια ενιαία αγορά που θα διέπεται από κοινού κανόνε για τι ε, διαδικτυακέ αγορέ και τι διαδικτυακέ ε, και τι μη διαδικτυακέ. Πιστεύω ότι στην αντίθετη περίπτωση απλά θα ενισχύσουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Εξού και το ζήτημα της ε, αποτελεσματικότητας της πρότασης και ο κίνδυνος περιπλοκής των πραγμάτων αντί διευκολυνσής τους. Οι νέοι κανόνες οδηγούν σε νέους κοινού κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Περισσότερη πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα με χαμηλότερο κόστος αλλά με ισχυρότερη προστασία. οι συμβατικέ σχέσεις πρέπει να είναι ισορροπημένε με ενισχυμένη προστασία αλλά χωρίς επιπλέον άχθος για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάουταλα. Θα ήθελα να σχολιάσει. Ναι, είμαι λίγο περίεργη να κάνω μια ερώτηση συγκεκριμένα για αυτή την ιδέα ότι αναζητούμε μια έξυπνη λύση για το πώ οι συμβάσει θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο που να σχετίζεται με τη διάρκεια ζωή ε, και τι προσδοκίε των καταναλωτών. Ε, να ρωτήσω την Κομισιόν. Ναι, Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν. Να πω κάτι εν συντομία για τρία σημεία που αναφέρθηκαν από πολλού ε, βουλευτέ, Αλλά το πρώτο που θέλω να αναφέρω το σημείο που έθεσε η κυρία Χαταλά, το ζήτημα της διάρκεια ζωής ενός προϊόντος η βιωσιμότητα είναι κάτι που παίρνουμε σοβαρά στην Κομισιόν. Μόλις οδετήσαμε ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να επιτυχούμε είναι ε, προϊόντα μεγαλύτερης διαρκές ζωής. Το ζήτημα είναι πώς. Θεωρούμε ότι ε, συγκεκριμένη νομοθεσία για συγκεκριμένα προϊόντα είναι ο καλύτερος τρόπος να σας εξηγήσω γιατί. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας ηλεκτρικής σκούπας. Όταν την αγοράζουμε υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού και της σχετικής οδηγίας που λέει ότι πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει η ηλεκτρική σκούπα για 5.000 ώρες. Αν δημιουργηθεί και ένα όριο στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας για τις πωλήσει θα καλύπτεται με τη μία μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. αν, σε, στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων έχει συχνότητα και η ένταση χρήση. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει τη σκούπα για δύο χρόνια, αλλά αν τη χρησιμοποιεί σπάνια, θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά από τα δύο χρόνια. Αν τη χρησιμοποιεί κάποιο εντατικά, μπορεί να πάψει να λειτουργεί μετά από ένα χρόνο. Αυτό που λέω κατά βάση και η προσέγγιση που έχει επιλέξει η Κομισιόν είναι η εξή. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωή, σα φτιάξουμε ειδική νομοθεσία για συγκεκριμένα προϊόντα που θα αξιολογεί τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήση. Ενώ για το δίκαιο πωλήσεων έχουμε μία ενιαία λύση για όλε τι περιπτώσει που καλύπτει τεράστια ποικιλία πολλών διαφορετικών προϊόντων. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω, εν συντομία, το ανέφεραν πολλοί βουλευτέ, είναι το ζήτημα τη πλήρου εναρμόνιση. Η Κομισιόν έκανε μία πρόταση πλήρου εναρμόνιση γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της πλήρους εναρμόνευσης επιτυχάνουμε τους δύο στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Πρώτος είναι ότι οι πολιτές, ειδικότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουν ένα σύνολο κανόνων βάσει του οποίου θα μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την αγορά. Εάν υπάρχει μια ελάχιστη εναρμόνιση ή μια πλήρη εναρμόνιση συνδυασμένη με στοιχεία ε, ελάχιστης εναρμόνισης, θα πρέπει πάλι να ελέγχουμε τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη στα σημεία που έχουν εναρμονιστεί λιγότερο και αυτό συνεπάγεται δαπάνε. Και έτσι δεν θα επιτύχουμε το στόχο. Ο δεύτερο στόχο είναι να επιτύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία των καταναλωτών, ώστε οι καταναλωτέ να εμπιστεύονται τι ε, αγορέ στο εξωτερικό. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι πού θα βάλουμε τον πύχη. Το πρόβλημα είναι το κατά πώ θα γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι υπάρχει ένας ενιαίος πύχης ώστε να μπορούν με αυτοπίτηση να πάνε στο εξωτερικό και να πούνε ξέρω, ποιον, ποιο, ξέρω ποιος είναι ο πύχης, είναι εύλογη η προστασία. Οπότε εμεί θεωρούμε ότι η πλήρης εναρμόνιση θα επιτύχει τους στόχους ή ένα σύστημα ε, ε πλήρους εναρμόνισης σε συνδυασμό με ελάχιστη εναρμόνιση ή ελάχιστη εναρμόνιση δεν θα επιτύχει το στόχο. Και το τελευταίο που ήθελα να δείξω, που έθιξαν πολλοί βουλευτές είναι που βάζουμε το όριο μεταξύ των δύο προτάσεων του ψηφιακού περιεχομένου και των ε, διαδικτυακών πωλήσεων. Ναι, συμφωνούμε, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, δεν λέμε ότι το προτείναμε εμεί, αλλά ε, ο νομοθέτης φυσικά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η διάκριση θα πρέπει να αφησίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλίζει μια προσέγγιση που θα μας καλύπτει και στο μέλλον και δεύτερον, μια διάκριση που να είναι πρακτική, εφαρμόσιμη. Έχουν συζητηθεί πολλές προσεγγίσεις. Να αναφέρω μία που έχει συζητηθεί, το πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι αγοράσετε ένα πλυντήριο, πατάτε το start και δεν λειτουργεί. Η βλάβη θα μπορούσε να είναι στο λογισμικό ή σε ένα μηχανικό εξάρτημα του πλυντηρίου. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να το γνωρίζει. Έχει τρόπο να το γνωρίζει του πείτε ότι υπάρχει, αν πούμε ότι υπάρχει διάκριση ε, στο πού βρίσκεται η βλάβη, ο, ο καταναλωτή θα πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκεται το πρόβλημα, πού βρίσκεται η βλάβη, ώστε να ξέρει πού να αποταθεί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ε, ίσως για ένα πλυντήριο να μπορεί να το βρει ο καταναλωτή, αλλά στην περίπτωση μια τηλεόραση είναι αδύνατον. Οπότε, κατά βάση αυτό που συνιστούμε είναι να είμαστε κάπως προσεκτικοί γιατί ε, Κάποιε προσεγγίσεις που φαίνονται εύκολε όσον αφορά τη διάκριση ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα περίπλοκε στην πράξη. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να μας καλύπτει και στο μέλλον, δηλαδή να ταιριάζει στις σημερινές συνθήκες αλλά και οι συνθήκες που θα επικρατούν ε, στην επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία γιατί το διαδίκτυο των πραγμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται και οι οικιακές συσκευέ που θα έχουν θα περιλαμβάνουν λογισμικό το οποίο θα είναι προσπελάσιμο από το διαδίκτυο, θα αυξηθούν γεωμετρικά. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση που να μα καλύπτει όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τους ευρωβουλευτές για να βρούμε μια τέτοια λύση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο ή θα ήθελε η κυρία Χάτολα να πει κάτι. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, προσέθεσε το θέμα του REFIT. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Σλοβακική Προεδρία ε, πρέπει πράγμα να προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα με αυτή την οδηγία περί ενσώματων αγαθών για να υπάρξει και κάποια εναρμόνιση. Επίσης ε, προγραμματίζουμε μία μελέτη για τη σχέση ανάμεσα στα tangible goods, τα ενσώματα αγαθά και το equal design όχι equal, eco-design και οικολογικός δηλαδή σχεδιασμός. Μιλάμε για προϊόντα τα οποία υπολείπονται κατά πολύ των ε, ε, αιτιολογημένων προσδιοκιών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, with the kind permission of Mrs. <clears throat> Um, Regner, could we, uh, could we take point 31 first? Ε, κυρία Ρέγνερ, μήπως uh, Θέλετε να περάσουμε στο 31 γιατί η κυρία Χάουταλα θέλει να φύγει, αλλά και εσείς θέλετε να φύγετε. Σε αυτή πάμε στο 30. Ανταλλαγή απόψεων, uh, αποκάλυψη ε, πληροφοριών, ε, μισό λεπτό, κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το φόρο εισοδήματο από συγκεκριμένε επιχειρήσει ή υποκαταστήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι που δεν μπορώ να το αναβάλω, αλλά και εγώ έχω ένα συγκεκριμένο προπολογισμό χρόνου και δεν θέλω να τον παραμπώ. Ε, θα τα πω σχετικά γρήγορα. Ε, Πήραμε στις 12 Απριλίου μια σχετική πρόταση όσον αφορά τις αναφορές αναχώρα και θέλω να πω το εξής επ' αυτού. Για μένα είναι πολύ σημαντικό στην Επιτροπή να αναφέρουμε ότι πρόκειται για την αλλαγή της οδηγίας περί λογιστικών προϋπολογισμών. Και πλέον ε, έχουμε εναρμονιστεί και με τους συναντέλφου της Επιτροπής ΕΚΟΝ η φορολογική διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι επιχειρήσεις το χρωστάνε αυτό όχι μόνο στις φορολογικές αρχές ε, και στις ε, στα κρατικά ταμεία να ανταλλάσσουν δηλαδή αυτόματα πληροφορίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι η κοινή γνώμη έχει κάθε δικαίωμα να ενημερώνεται. Γιατί? Διότι τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες δεν προσφέρονται και δεν παρέχονται εν κενό, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την υποδομή, δηλαδή τους υπαλλήλους, άρα οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενημερώνονται στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται. Σας λέω, είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε εν κενό. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε επί της έκθεσης τάξε όπου ξεκαθαρίστηκαν κάποια θέματα. Η Ολομέλεια δηλαδή επέκρινε δρυμύτατα ότι η πρόταση της Κομισιόν της 12ης ε, Απριλίου ε, υπολείπεται στα κριτήρια, στο πεδίο εφαρμογής, όπως επίσης και στα, στις τιμές, στο επίπεδο κατόφλι για την υποχρέωση ενημέρωσης. Θα αναφερθώ στους τρεις αυτούς τομείς, αλλά όπως σας είπα γνωρίζω πολύ καλά το, μέχρι που έχουμε προχωρήσει σήμερα. 150 εκατομμύρια, αυτό είναι το ε, κατώτατο όριο και θέλω να σας πω ότι βεβαίως και έχω μεγάλη κατανόηση για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια εναρμόνιση με το BEPS, την οδηγία περί BEPS και θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι γνωρίζουμε και άλλες ε, τιμές ε, κατόφλι στην προηγούμενη οδηγία, για, στην προηγούμενη θητεία μιλήσαμε για τις οδηγίες που αφορούν στην εξόριξη μεταλλευμάτων και είχαμε και την οδηγία των ε, ε, μετόχων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη του οι σκιώδεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεπής προσέγγιση. Δεύτερον, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογή. σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επίσημα έκθεση ανά χώρα, αλλά έχει έκθεση ε, κράτη-μέλη ανακράτη-μέλη, κράτη-μέλη, συν φορολογική παράδοση. Δηλαδή η Κομισιόν αναφέρεται περισσότερο στο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να αποκτήσει η Κομισιόν συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό για μένα είναι ένα χάσμα, ένα κενό ε, και γι' αυτό ε, δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει η Κομισιόν. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι όταν δεν τηρείται και δεν εφαρμόζεται η οδηγία, θα πρέπει κάτι να πούμε για τις κυρώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα Swiss Leaks, στα Panama Papers υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και εμείς ε, ως ε, βουλευτές προσιλωμένοι και δεσμευμένοι απέναντι στην αλήθεια, αυτά δεν μπορούσαμε να τα αποκτήσουμε διαφορετικά. Άρα δηλαδή φέρουμε ευθύνη έναντι των πολιτών της Ευρώπης ε, ε, με νύχια και με δόντια να επιτύχουμε αυτές τις εκθέσεις αναχώρα. Ε, πολύ γρήγορα τα από αυτά τρέχοντα. Ήταν έτσι μια δική μου πρώτη προσπάθεια για να υπάρχει και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίω για μένα είναι πολύ σημαντικό με του σκιώδει ηγητέ να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία και κατόπιν του κλείνοντα, ε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ λιγάκι και στο χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, για το καλοκαίρι. Προβλέπετε να εργαστούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις 12-13 Οκτωβρίου να υποβάλουμε την έκθεση. Λίγο πολύ δηλαδή ήδη το Σεπτέμβρη να δοθεί έκθεση για μετάφραση. Και κατόπιν η, η διορία είναι 27 Οκτωβρίου για τις τροπολογίες προφανώς και ε, και μετά, έκτοτε δηλαδή, ε, να δουλέψουμε πολύ γρήγορα ε, για να φτάσουμε στην ψηφοφορία σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, πάρα πολύ γρήγορα αυτά είχα να πω για τις εκθέσεις αναχώρα. Ευχαριστώ κύριε Ε Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ του συναδέλφου Καρίν που εκπροσωπώ, θέλω να συγχαρώ την κυρία Ρέγκνερ και να πω ότι η ομάδα ECR υποστηρίζει την έκθεση αυτή μετά το σκάνδαλο LuxLeaks. Θεωρούμε ότι είναι καλή αυτή η πρόταση. Από τη στιγμή που θέλει να υπάρχει αποκάλυψη πληροφοριών και κυρίως στοχεύει στις πολυεθνικές. Βέβαια, η διεύρυνση του παιδί εφαρμογή, δηλαδή να καλύπτονται και οι ΜΜΕ, είναι πολύ μεγάλο άχθος Θεωρούμε επίσης ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής της πρότασης αυτής. Χωρίς όμως να βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα απέναντι σε τρίτες χώρες. Να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε συναρπαστικές συζητήσεις και να ξέρουμε ότι οι τρίτες χώρες δεν θέλουν να ξεπεράσουν τους κανόνες του ΩΣΑ. Ευχαριστώ. Κύριε Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρίγνερ, την εισηγητριά μας, για την εισήγησή της. Εγώ θα κάνω κάποιες ε, γενικέ φύσεως παρατηρήσεις, γιατί για τις λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κατά τους επόμενους μήνες. Μετά λοιπόν ε, τις δημοσιεύσεις ε, των προηγούμενων μηνών, Panama Papers ε, και Swiss Leaks, τίθενται ορισμένα σημαντικά θέματα και ε, ρωτώ, επιθυμούμε να κλείσουν τα φορολογικά κενά, επιθυμούμε να πάψει να υπάρχει η φοροαποφυγή. Θέλουμε κάποια στιγμή πραγματικά οι φόροι να ε, καταβάλλονται στο χώρο όπου προκύπτει η προστιθέμενη αξία και αν ναι, αυτό πώς θα το πετύχουμε. Η διαφάνεια είναι σωστός δρόμος και αν όχι, τι είδους εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν. Κυρία Ρίγνερ, αναφερθήκατε στην έκθεση τάξε 2, επί της οποίας ε, ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια Σήμερα συστήθηκε ε, ε, επιτροπή για τα Panama Papers. Αυτά όλα πρέπει να τα απαντήσουμε. Και νομίζω ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι όσον αφορά το θέμα της φοροαποφυγής και των φορολογικών κενών, το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστεί επί των θεμάτων αυτών. Και μια γενική φύσεως παρατήρηση, γιατί νομίζω ότι όσον αφορά τη φοροαποφυγή θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα αν τα κράτη-μέλη είχαν επιτύχει να υπάρξει μια ενιαία φορολογική βάση. Ε, αυτό είναι εκείνο, ή ενοποιημένη μάλλον, ενοποιημένη φορολογική βάση. Αυτό είναι εκείνο το οποίο με απασχολεί, το πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ε, περάσουμε σε νομοθετήματα. Αν υπήρχε αυτή η ενοποιημένη φορολογική βάση, τότε θα ήμασταν και σε θέση να επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση φορολογικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Τα λέω αυτά έχουν κατά νου και το Brexit. Ε, όλα αυτά ε, συνέβησαν όχι γιατί δεν υπάρχει ε, η βούληση από τα κράτη-μέλη. Αν εμείς είχαμε λειτουργήσει περισσότερο προληπτικά θα είχαμε αποφύγει πολλά πράγματα. Επανέρχομαι στην πρόταση. Καλό που την υπέ... υπέβαλε η Κομισιόν λεπτομέρειες θα συζητηθούν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους ε, που πρότεινε στους σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουν για να διαπιστώσουν κατά πόσο μπορούν να καταλήξουν σε μια συμβαστική πρόταση. Για μένα είναι σημαντικό τις προτάσεις του ΩΣΑ από το πρόγραμμα δράσης ε, BEPS ε, να μην τις αντιπαραβάλλουμε με αυτό το πρόγραμμα γιατί νομίζω ότι εμείς φέρουμε ευθύνη για τις επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη να ανταγωνίζονται επί ίσων όρων και όχι να εγκρίνουμε κάτι το οποίο όπως σας είπα αντιπαρατίθεται στους κανόνες του ΩΣΑ. Επίσης το βρίσκω πολύ καλό ότι επιχειρήσεις που δεν έχουν πηγατρικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριληφθούν και αυτές γιατί μόνο έτσι θα επιτύχουμε πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού. 750 εκατομμύρια ευρώ, αυτή η τιμή κατόφλη, καλό είναι αυτό. Και αυτό για να μπορέσουμε να είμαστε και συνεπείς με τους κανόνες του ΟΣΑ. Άκουσα τι είπατε σε σχέση με άλλες οδηγίες, κυρίως σε σχέση με την οδηγία περί μετόχων. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Και επίσης και το άρθρο 48 σε δύο κατάλογος αν νομίζω εκεί γίνεται λόγος ε, για τις ε, πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις ε, να δούμε κατά πόσον αυτό είναι λογικό για να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι επιχειρήσεις μας πράγματι δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση αυτά εν είδη πρώτης τοποθέτησής μου κυρία εισηγήτρια και έχω και άλλη μια ερώτηση, γιατί έτσι δεν είμαι καλά ενημερωμένη. Το θέμα της σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την ΕΚΟΝ έχει ρυθμιστεί αυτό και αν ναι, πάνω σε ποια βάση. Τι διαδικασία θα εφαρμόσουμε, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις. Δεν το έχετε εξαντλήσει το θέμα, από ό,τι βλέπω νεύεται αρνητικά, άρα δηλαδή το θέμα συζητιέται ακόμα, κατόπιν τούτου καλύφθηκα στην ερώτησή μου. Ευχαριστούμε. Αυτή η σύγκρουση αρμοδιοτήτων ε, δεν έχει ακόμα επιλυθεί. επιληθεί. Θα ασχοληθούμε με αυτήν ε, μέσω διαμεσολάβησης με την κύριο Μπούζεκ. Θέλει να σχολιάσει κυρία Ρέγνερ. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να κάνουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Το θέμα των αρμοδιοτήτων ε, δίσταζε λιγάκι γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και ε, χιλιάδες χρόνια. Το θέμα είναι σημαντικό, να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας, ε, αυτά που είπατε επί του περιεχομένου και προσβλέπω στη συνεργασία. Θα ήθελε η Κομισιόν να πει κάτι. Α, η κυρία Βίξτρεμ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, παρότι ήρθα τελευταία. Οι εκθέσεις κατά χώρα είναι ιδιαίτερα προσφυλής, το ίδιο και στην ομάδα μου. Ασχοληθήκαμε με αυτές στην εκθέση Κοφεράτη και θυμάμαι συναρπαστικές συζητήσεις επί του θέματος. Τώρα που έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν επί του θέματος, αυτό πρέπει να μας χαροποιεί αρμόζει πιστεύω στο πλαίσιο αυτό να ασχοληθούμε με τις εκθέσεις κατά χώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό αποτελεί προσδοκία των πολιτών. Θέλουν οι πολίτες μας να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τις απάτες και τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης όποια συμβαίνουν. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε αυτό το ζήτημα να το ρευνήσουμε σοβαρά και επίσης και η σπουδαιότητα της διαφάνειας θα κάνει τον κόσμο να νιώσει άνετα, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να τα διασφαλίσουμε όλα αυτά. 75% σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Ιουνίου φέτος λένε ότι θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερη δράση. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Είναι υποχρέωσή μα πλέον, ωστόσο έχω κάποιε αμφιβολίε για το πόσο αποτελεσματική θα είναι μια μαύρη λίστα μη συνεργάσιμων φορολογικών αρχών. Ενδεχομένως ο τραπεζικός τομέας, η υλοτομία, ε, ο τομέας των μεταλλίων να είναι κάπως διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά αν μπορούμε να έχουμε τέτοια ε, ε, τέτοιες αναφορές, ε, εκθέσει κατά χώρα σε διάφορου τομεί, γιατί να μην έχουμε και εδώ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία. Επειδή η πρόθεση της Κομισιόν εξαιρεί 85 έως 90% των πολυεθνικών αυτό παγκοσμίως, αυτό μας δημιουργεί κάποιο προβληματάκι. Και δεν υπερβάλλω. Εγώ αναμένω να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους και ελπίζω να βρούμε τελικά μια ισχυρή κοινή θέση και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην ε, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Είστε ευπρόσδεκτοι. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη δήλωση κομισιών επειδή τελειώνει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με την πρόταση της Κομισιόν που είναι ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και φυσικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε την αποφυγή θα συνεργαστούμε με την εισηγητρία, του Σκιώδη και το Κοινοβούλιο. Να σα πούμε επίση ότι το Συμβούλιο Σημειονίδη Πρόοδο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση τη πρόταση επί ε, Δανέζικη Προεδρία. Επί συγγνώμη, Ολλανδική Προεδρία και η Σλοβακική Προεδρία θα συνεχίσει πέντε τη σκητάλη. Άρα, καλά κάντε και εσεί και ξεκινάτε τώρα την ε, εργασία σα επ' αυτού. Σε ό,τι αφορά ε, τα κατόφλια ετέθη το ερώτημα. Θέλω να σας πω ότι το κατόφλι το οποίο επιλέξαμε αντικατοπτρίζει αφενός την ανάγκη να μην επιβαρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις με αυτό το διοικητικό φόρτο. Επιλέξαμε λοιπόν με αυτή την πρόταση 750 εκατομμύρια 10% των, των ε, πολυεθνικών, 6.000 περιπετέρειε δηλαδή υπόκειται σε αυτή την υποχρέωση. Το 10% αυτών των πολυεθνικών όμω είναι το 90% του τζίρου των πολυεθνικών. Σε αυτό το ποσό αντιστοιχεί. Άρα νομίζω ότι πολύ καλά επιλέξαμε αυτό το ποσοστό και φυσικά είμαστε ανοιχτοί να συστήσουμε το Κοινοβούλιο και αυτό και όλα τα άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ για τη σημαντική αυτή επεξήγηση. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο τη μερική διάταξη και δεν μπορούμε να συζητήσουμε το 31, δεν είναι η συγκεντρία μαζί μας πια. Έφυγε η κυρία Χάουταλα, οπότε θα πάμε στο σημείο 32. Ανταλλαγή απόψεων για μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Το λόγο έχει η συγγήτρια η κυρία Κομοντίνη. Okay. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά βάση πολύ σύντομη αυτή η έκθεση. Βέβαια, ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δημιουργικός και πολιτισμικός κλάδος δεν ε, ε, αξιοποιούνται πλήρως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κατακαιρματισμό και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Για το νέο πρόγραμμα το επιχείρημα είναι ότι η δημιουργική πολιτισμική κλάδη παρά το δυναμικό τους ε, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο δεν αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς ιδίως λόγω όπως είπα του μεγάλου κατακαιρματισμού. Επίσης ε, το νέο πρόγραμμα Creative Europe ζητεί ενίσχυση ε, της προσαρμογής των δημιουργικών πολιτισμικών κλάδων στην παγκοσμιοποίηση. Πιο στοχευμένη εστίαση στη διακρατή υποχρεωτική κυκλοφορία έργων. Θα οδηγήσει σε πιο πολλέ εμπορικέ συναλλαγέ εντό τη εσωτερική αγορά, περισσότερο εθνέ εμπόριο, θα αυξήσει και τα έσοδα των τομέων αυτών. Επομένω, ποιο είναι το πεδίο, ποια είναι, ποιο είναι το κόνσεπτ. Ε, είναι ευρύ και περιλαμβάνει τις ε, καστικές τέχνες, ε, τις... τα βιντεοπαιχνίδια, τα νέα μέσα, αρχιτεκτονική αρχιτεκτονική, διαφήμιση, eco και πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχουν όμως κοινά θέματα για όλους αυτούς τους τομείς. Κάποιοι βέβαια, κλάδοι, έχουν κάποια μεμονωμένα χαρακτηριστικά, όλοι συνεισφέρουν όμως τη δημιουργία θέσεων εργασίας και έχουμε και τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων. Η δημιουργικότητα πρέπει να τονωθεί σε όλου του τομεί τη οικονομία, με υπηρεσίε που θα ενισχύουν την αλυσίδα τη καινοτομία και θα προσφέρουν πρόσβαση σε όλε τι μορφέ στήριξη τη καινοτομία. Μια από τι βασικέ προκλήσει είναι να δημιουργηθούν προποθέσει για επενδύσεις ε, στη δυναμικότητα των τομέων αυτών, να βρουν διασυνοριακά ένα άλλο, ένας άλλος διάβλος είναι να στηριχθεί καινοτόμως επιχειρηματικότητα και με βάση την κρίση την πρόσφατη πιστεύω ότι οι δύο σημεία πρέπει να προσαρμοστούν ίσως και να επανεξετάσουν συνολικά την προσέγγισή τους. Γι' αυτό απαιτείται ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τις ΜΜΕ, θα τις καθοδηγεί, θα βελτιώνει την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, θα μεγαλώνει τις δυνατότητες τους για καινοτομία και θα προωθεί το καινοτόμο επιχειρηματικό πνεύμα. Κάποιες από τις προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ανάγκη ανάπτυξη συνεκτική μακροπρόθεσμη βιομηχανική ε, στρατηγική, προώθηση πολιτισμικών και δημιουργικών κλάδων ω προτεραιότητα σε όλε τι πολιτικέ τη Ένωση. Επίση, το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί για την αλυσίδα στην ψηφιακή εποχή, ώστε να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε αυτών των κλάδων και να οδηγεί σε βελτίωση των αμοιβών των δημιουργών. Έχουμε και τη μεταρρύθμιση στο δικαίωμα του δημιουργού για να βρεθούν κατάλληλε λύσει για του κατόχου δικαιωμάτων καταναλωτέ δημιουργού. Έχουμε εξαιρέσεις όμως ευθύνη μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι για τις υπηρεσίες που προωθούν το περιεχόμενο. Σήμερα καταναλώνεται πολύ περισσότερο δημιουργικό περιεχόμενο από ό,τι παλιά πλατφόρμες ε, μεταφόρτωσης περιεχομένου, αναπτύσσονται κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε συγκριτικό, συγκριτική αύξηση των εσόδων των παραγωγών με την αύξηση της κατανάλωσης. Υπάρχει ένα κενό ε, αξίας. Δεν το παίρνουν το κέρδος η παραγωγή και η δημιουργή. Υπάρχει μια αθέμητη αγορά και έτσι τίθεται και ε, σε κίνδυνο η ενία αυτή αγορά για τους πολιτισμικούς δημιουργικούς κλάδους. Το χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο έκθεσης και για την κατάσταση τροπολογιών, τουλάχιστον μάλλον για την σύνταξη της έκθεσης, είναι πολύ σύντομο. Για την κατάσταση τροπολογιών προτείνεται ως προθεσμία από τη Γραμματεία 6 Σεπτεμβρίου. Και για την εξέταση τροπολογιών και συμβαστικών τροπολογιών προτείνεται ο Οκτώβρης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε συναντήσεις με τους σκιώδες μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Και η ψηφοφορία προβλέπεται για τον Δεκέμβριο. Δεν έχει βεβαιωθεί ακόμη προθεσμία. Ε, στην Ολομέλεια μάλλον για τον Δεκέμβριο πάντως ε, πηγαίνουμε. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τι θέλουν να πούν οι σκιώδες ηγητές και φυσικά θα συνεργαστώ μαζί τους. Ευχαριστούμε κύριο Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ και χρόνια γνωρίζαμε ότι ο πολιτιστικός τομέας δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Εγώ στις δικές μου εκθέσεις που έχω συντάξει έχω υπερασπιστεί τα δικαιώματα δημιουργού δημιουργού και ανέκαθεν ήμουν υπέρ της ε, αμοιβή των δημιουργών. Αλλά ο τομέας αυτός είναι πολύ πιο ευρύς. Οι ε, πολιτιστικοί τομής ε, τονώνουν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και συμμετέχουν στην παιδεία, στην αστική πολιτική και σε άλλες πολιτικές. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά σε εθνικό επίπεδο. Εδώ το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την ενημέρωση βέλτιστων πρακτικών ή να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που χρειάζονται τη βοήθειά μας ώστε να εκπονήσουν τη δική τους ε, νομοθεσία. Πιστεύω ότι ε, μια εναρμονισμένη πολιτική δεν είναι καλή ιδέα για το θέμα αυτό. Η αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Αλλά δεν πάει να είναι και ασταθής και δυναμική. Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά, τα κράτη-μέλη και οι δήμοι ε, πρέπει να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές και τις χρηματοδοτήσεις. Δύο πρέπει να κερδίσουν, η δημιουργή και η δημιουργική βιομηχανία. Ε, Mr. Κύριος Νεγκρέσκου, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εστιαστούμε, πιστεύω, στις ε, νομικές πτυχές του εγγράφου. Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε θετικά στο εγγραφό και πρέπει να υπογραμμίσουμε λίγο περισσότερο την ανάγκη ύπαρξη ενός κοινού νομικού πλαισίου όταν μιλάμε για τον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα, όχι μόνο τη βιομηχανία. Αναφέρομαι σε αυτό στο τομέα, γιατί είναι πιο ευρία η έννοια από το είναι η βιομηχανία. Αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να αναφερθούμε και σε όλε τι πτυχέ και τα προβλήματα που σχετίζονται με τον τομέα αυτών. Δεύτερον, πιστεύω πρέπει να καθορίσουμε την πολιτισμική και δημιουργική βιομηχανία ή τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, γιατί νοείται με διαφορετικού τρόπου ε, σε διάφορα μέρη τη Ευρώπη. Οπότε πρέπει να μα απασχολήσει και αυτό. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο για την ε, αλυσίδα αξιών, ειδικότερα στο σημερινό πλαίσιο όπως αναφέρει ο εισηγητής, αλλά ταυτόχρονα, συγγνώμη, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ε, προστατεύσουμε τους δημιουργούς ε, από την παραποίηση. Πρέπει να το αναφέρουμε σαφώς στην εκτίση και να προστατεύσουμε φυσικά τον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση εξορροπώντας ε, τους παρόχους με τους δημιουργούς ε, και τους καταναλωτές, ώστε όλοι να κερδίζουν από αυτό το παιχνίδι. Ο τομέας αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σημαντικό διότι όλοι αυτοί οι φορεί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τον οποίο πρέπει να καθορίσουμε εμεί και να βεβαιωθούμε ότι θα βελτιωθεί η αμοιβή για όλου, αλλά κυρίω για του ε, ε, δημιουργός ε, κατά την απόψή μου. Τέλος, εξίσου σημαντικό, πρέπει να κάνουμε κάτι για την επιχειρηματικότητα στον τομέα αυτό, να δώσουμε κίνητρα για τις μικρές επιχειρήσεις, να τους βοηθήσουμε, να τονώσουν τις δραστηριότητε τους. Είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε, να κάνουμε κάτι που θα βοηθήσει τα κρατημένα να αναπτύξουν περαιτέρω τον τομέα αυτόν. Και τέλος, δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε την αγορά να οδηγήσει τις εξελίξεις. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους, τους δημιουργούς να δείξουν τις εξελίξεις. Θα τα βρείτε αυτά στις τροπολογίες που θα υποβάλει ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Σκέστερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την κυρία Κομοντίνη για την έκθεσή της. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να υπάρχει μια συνεπής ενωσιακή πολιτική για τον ε, πολιτισμό και για τον δημιουργικό κλάδο, να μεριμνήσουμε ότι ώστε η δημιουργή να είναι η καρδιά του πολιτισμού. Και πρέπει να είναι σαφές ότι κυρίως ε, οι δημιουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι την εποχή της ε, ψηφιοποίησης πολλές φορές είναι οι χαμένοι. Μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, πολλοί εξ αυτών επιθυμούν να έχουν ε, θέσεις ε, ασφαλισμένες και επιθυμούν να έχουν και κάποια προοπτική σε προχωρημένη ηλικία, να μπορούν να απολάβουν τότε κοινωνική ασφάλιση. Για να το επιτύχουμε αυτό, ε, πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα του πώς οι δημιουργοί στις διαπραγματεύσεις τους αυτές που διεξάγουν να ενισχυθούν στη διεκδίκηση των ε, δικαιωμάτων τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, τις ε, εταιρείε αυτές που θα διαπραγματεύονται τα δικαιώματά του συλλογικά είναι πολύ σημαντικές αυτές και μέσω αυτών ίσως ε, οι δημιουργοί να μπορούν να διαπραγματεύονται ίσης όρης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι σε αυτή την αλυσίδα προστέμενης αξίας χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, κυρίως στον μουσικό κλάδο. Γιατί σε τελική ανάλυση και η μουσική μπορούν να παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία. Άρα δηλαδή που καταλήγουμε, καταλήγουμε σε αναδιανομή από τους μεγάλους παίκτες, YouTube ας πούμε, στους ε, καλλιτέχνες, στους μεμονωμένους, κάπως να βρεθεί ένα σύστημα για να υλοποιηθούν οι στόχοι μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό το να υπάρχει συνεπής πολιτική και όλα αυτά κάτω από το εξής light motif. Το light motif θα μπορούσε να είναι ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και παράλληλα δίκαιη αμοιβή και αποζημίωση για τους δημιουργούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Θέλει τίποτα η συγγήτρια. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι άκουσα σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου και νομίζω ότι λίγο πολύ τα ίδια σκεπτόμετα και γι' αυτό ε, χαίρομαι. Προσβλέπω συνεργασία με κάθε ένα εξ αυτών. Έκλεισε και αυτό το θέμα, λέει ο Πρόεδρος, και πάμε τώρα στο υπαριθμό 33, στο 33, που είναι η έκθεση αποστολής ε, μετά την επίσκεψη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στη Γεωργία από τις 29 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η αντιπροσωπεία μας δεν θα έλεγα ότι ήταν πολυάθμη Μπρεξερών, Χάουταλα, και ο υποφαινόμενος. Και ο υποφαινόμενος λοιπόν συμμετείχαμε σε αυτή την επίσκεψη διάρκειας δύο ημερών και διαπιστώσαμε ότι η Γεωργία σημειώνει σημαντική πρόοδο στην, ε, στη μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού συστήματος. προβλέπουν πλέον νέους ε, θεσμούς και τα προβλήματα που προκύπτουν έχουν σχέση με την εφαρμογή. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η κατεύθυνση που λαμβάνει η γεωργία είναι σωστή. Να σας αναφέρω απλώς ένα σύντομο κατάλογο θεσμών με τους οποίους συναντηθήκαμε, χωρίς ονόματα βέβαια, με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, με τον επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Monitoring της Γεωργίας, τον πρόεδρο της Βουλής, ε, τον ε, Ombudsman, τον διαμεσολογητή ε, με πολλούς της κοινωνίας των, πολιτιών, κοινωνίας των πολιτών, Euronest. Επίσης συναντηθήκαμε με τον ε, επικεφαλής ε, της αντιπολίτευσης, ε, των μειονοτήτων, τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Επικρατείας της Γεωργίας για την ένταξη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωατλαντική της ενσωμάτωση. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις. Αν όχι, τότε πάμε στο 34 παρακαλώ παρουσίαση του αποτελέσματος της ε, αποστολής ε, στο Πεκίνο, στην Κίνα και ο κύριος Τζαμπάσκι θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία γιατί οργάνωσε πολύ καλά αυτή την επίσκεψη και δεν ήταν καθόλου εύκολο καθότι οι κινέζικες αρχές δεν επέδειξαν ιδιαίτερη ευελιξία. Μπορώ να πω εν γέννη πως Αυτοί που μας κάλεσαν ε, επέδειξαν ιδιαίτερη φιλοξένη. Όχι όμως και τόση ευελιξία σε ό,τι αφορά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς για την Κίνα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την ε, οργάνωση χρονικά της επίσκεψης αυτής. Η Κίνα όπως ξέρετε, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις απομιμήσεις και παραποίησεις προϊόντων. Στο ξενοδοχείο μας, ε, μέχρι και εκεί, ε, είχαμε πρόβλημα με τα πλαστά χαρτονομίσματα, να φανταστείτε. Τέλο πάντων, εμεί θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τι κινέζικε αρχέ. Επιβεβαίωσαν και οι ίδιε την δική του προθυμία για να συνεργαστούν με εμά. Θα πρέπει να δούμε και να εργαστούμε από κοινού για να κλείσουν ε, τα εργαστήρια, επιχειρήσεις που πλαστογραφούν ε, νομίσματα για παράδειγμα. Επίσης, ζητήσαμε να υπάρξει πολύ περισσότερη συνεργασία σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Και αρχές ήθελα να συζητήσουμε για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, η Επιτροπή μας δεν είναι ε, ο καλύτερος ε, συνομιλητής, δεν είναι ο πιο συνομιλητή για αυτά τα θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τη Γραμματή για μια ακόμη φορά και την κυρία Κομοντίνη επίσης θέλω να ευχαριστήσω και για τις διαπραγματεύσεις ε, και τη διπλωματικότητα που επέδειξε σε μια κατάσταση που δεν ήταν και τόσο εύκολη. Ευχαριστώ κύριε Κομοντίνε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι την προσωπία αυτή ήταν πολύ καλή. Είχαμε συναντήσει με διάφορους εκπροσώπους και εξωματούχους από κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι είδαν και είδαμε και εμείς ότι υπήρχε ένα πολύ σεφές πρωτόκολλο το είδαμε όλοι, σε όλες τις συναντήσεις μας ήμασταν όμως ευέλικτοι, ανοιχτοί στα ερωτήματα, παρέχαμε πληροφορίες, όμως πάντοτε ή συχνά τέλο πάντων ε, είχαμε ε, απέναντί μας ε, αξιωματούχους σε δεταγμένη υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν ε, κάποια ζητήματα που θέλαμε να αναφέρουμε σημαντικά σε ό,τι αφορά το διάλογο με την Κίνα, τα είπε και η κοινή αντιπροσωπεία στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματο, στο Κογκρέσο, για να συζητήσω. Και ο Τζαμπάσκι είπε ότι είχαμε αυτό το ψήφισμα για τη χωρί καθεστώτο οικονομική αγορά στην Κίνα. Αυτό είχε κάποιε ανησυχίε. Νομίζω τι καθησυχάσαμε, τουλάχιστον τι εντάσει τι περιορίσαμε, λέγοντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε τηρεί τι ε, διεθνεί ε, υποχρεώσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, μετά την πρώτη μας συνάντηση με το Κογκρέσο δεν ε, ξανατέθηκε το θέμα αυτό και νομίζω ότι έγινε προσπάθεια να αποφευθεί ε, να τεθεί το θέμα αυτό και στις άλλες. Να τις πάντα παρακολουθήσει κάποιος από το Κογκρέσο, ε, από το συνέδριο μάλλον ε, του κόμματος, ε, όλες τις συναντήσεις της παρακολουθούσαν. Όπως είπα, λόγω τον προσπαθεί να εξαρτοποιηθεί περισσότερο το δικαστικό σώμα από το ε, κόμμα. Δεν έχουμε πετύχει και πολλά. Rule by law θα έλεγα ότι ισχύει. Δηλαδή κυβερνούν μέσω του δικαίου στην Κίνα. γίνονται κάποιες προσπάθειες για, το, για τις ποινικές διαδικασίες, για το δίκαιο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Βέβαια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γιατί συναντηθήκαμε με κάποιους επιχειρηματίες εκεί, αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό και εμπόδια σε ό,τι αφορά τι διοικητικέ διαδικασίε για την καταχώρησή τους ε, και επιβολή κάποιων ε, διατάξεων σε ό,τι αφορά ιδίω παραποίηση, πλαστογράφηση και πειρατεία καινοτομία και τεχνολογία. Είναι σημαντικό τομέα και για να τον πετύχουν, πετύχουν τους στόχους τους ακολουθούν μια επιθετική πολιτική οι Κινέζοι και αυτό συνάντησε την έντονη μας αντίσταση. Είπαμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στις δομές διαλόγου που έχουμε την Κίνα ώστε η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, IPR, δηλαδή πνευματικά δικαιώματα να προστατεύονται. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα επίση τι εξελίξει στην Κίνα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή εποχή, αν θέλουμε να προσαρμοστούμε μας είπαν ότι μπορούμε να αναμένουμε σύντομα αλλαγέ στην νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα που θα ε, προσαρμόσει ε, την Κίνα πιο πολύ στη νέα πραγματικότητα της ψυχικής εποχής. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη και τη δυναμική προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στην Κίνα. Είναι τελείως διαφορετική κατάσταση σε σχέση με το τι ισχύει εδώ. Και συχνά ε, εστιάζουμε στο υλικό, τα προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα ή παίρνουν την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και μετά αναπτύσσουν τα σχετικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη. Κυρία Άνιμπορ, και εγώ ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας και θα ήθελα να προσθέσω ότι και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές και την Τερέζα που ηγήθηκε της αντιπροσωπείας. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον διότι είναι μεταβατική η περίοδος, περνούν από μια κλειστή χώρα και οικονομία σε έναν πιο ανοιχτό κόσμο και προσπαθούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα όσα κάνουν. Ήταν δύσκολο λοιπόν, ξέρετε τις περισσότερες συναντήσεις δεν κάναμε ιδιαίτερα διάλογο, μας έλεγαν αυτό που θέλουν να μας πούν. Εμείς ε, προσπαθούσαμε κάπως να αποκριθούμε αλλά δεν ήταν αμφίδρομη η διαδικασία. Αλλά αυτό δεν υποβαθμίζει την ποιότητα της επαφής. Ήταν χρήσιμη γιατί όσο περισσότερο ανοιχτούμε προς αυτό, τόσο περισσότερο θα ανοιχτούν και αυτοί. Πιστεύω ότι έχει μια αξία δηλαδή με το δικό του τρόπο. Τέλος, ε, σημείο 35 έως 38 εξέταση των εκτελεστικών πράξεων και εκτελεστικών μέτρων και το λόγο έχει η συγγήτρια κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μένα για τα τελευταία τέσσερα θέματα ε, πρόκειται για τις κατεξότηση πράξεις και τα εφαρμοστικά μέτρα και μπορώ να σας αναφέρω μία ευχάριστη είδηση. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε όλα αυτά έτσι ώστε όλοι μας μπορούμε με την ησυχία μας όχι μόνο σήμερα να κλείσουμε τη συνεδρίαση αλλά και να πάμε στις ε, θερινές διακοπές. Και το λέω αυτό ε, γιατί όπως ε, σας είπα για μένα είναι η, τελευταία, η εξέταση των τελευταίων θεμάτων. Ευχαριστώ τον κύριο Γκριμάλτη και εύχομαι σε όλους σας καλές διακοπές. Επειδή Αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχουν ενστάσει, μπορούμε να κλείσουμε αυτά τα σημεία και το πρόγραμμα μας για τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ήθελα να σε ευχηθώ και εγώ ευχάριστες θερινές διακοπές και τα ξαναλέμε το Σεπτέμβριο.